Κυρίες, καθίστε. Κύριοι, euh, Λοιπόν, ε, σήμερα το πρωί έχουμε εδώ τον κύριο Κλάπενάουερ, ο οποίος είναι ο διευθυντής ε, της ε, μη στρατηγικής δυνατότητας σχεδιασμού και διεξαγωγής επιχειρήσεως και διοικητή των μη στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και μετά τον, ε, ε, τον εκπρόσωπο του ιδιαίτερου γραφείου του Γενικού Γραμματεία του ΝΑΤΟ και αν δεν υπάρχει αντίρρηση θα ήθελα να σας πω ότι 16 Οκτωβρίου θα έρθει ο κύριος Βέης από το Ευρωπαϊκό Γραφείο ε, Αμήνης. Πρόκειτο να συναντηθούμε και με τον Ναύαρχο ο Χάτσον ο οποίος ε, διευθύνει την επιχείρηση Αταλάντη αλλά ανεβλήθη η ημερομηνία αυτή γιατί συμπίπτει με μια άλλη συνεδρίαση και έτσι θα βρούμε μια άλλη ευκαιρία να δούμε τον κύριο Χάτσον προβλέψουμε να προβλέπουμε πριν το τέλος του χρόνου να επισκεφθούμε και το Γενικό Επιτελείο του ΝΑΤΟ και ε, θα ε, ε, θα ε, συναντηθούμε και μετά θα συζητήσουμε με τους συντονιστές για να συζητήσουμε για τις, για τα ταξίδια και τις αποστολέ στο εξωτερικό. Λοιπόν, χωρίς να χρονοτριβούμε, χαιρετίζω τον κύριο Κλόμπενχάουερ διευθυντή του CPCC ε, είναι μια σύνμηση την οποία σας παρακαλώ να μας διευκρινίσετε και επειδή υπάρχουν πολλά νέα μέλη καλό θα ήταν ε, να εξηγήσετε στους ευρωβουλευτές και εγώ συγκαταλέγομαι σε αυτούς ε, τι σημαίνει το CPCC και να αναφερθείτε στις ε, πολιτικές ε, επιχειρήσεις των οποίων υγείστε υπάρχουν δέκα τέτοιες επιχειρήσεις σε ενεξελίξη και ε, θα ήθελα για τα θέματα αυτά να μας τα παρουσιάσετε και στη συνέχεια ε, θα σας κάνουμε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ε, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να ενημερώσω την, υποεπιτροπή σας τόσο νωρίς με το ξεκίνημα του νέου κοινοβουλίου. Να σας πω κάποια ιστορικά στοιχεία για την μη στρατιωτική ΕΠΑ της οποίας είμαι υπεύθυνο. Κατόπιν θα δώσω μία γενικότερη εικόνα των ευρωπαϊκών αποστολών για τις οποίες είμαι υπεύθυνο και θα δώσω έμφαση στις τρεις σημαντικότερες κατά την άποψή μου το Αφγανιστάν, το Κωσυφοπέδιο και την Γεωργία. Αφήνοντας τις υπόλοιπες αποστολές για τις οποίες μπορούμε να επανέλθουμε αν θέλετε. Θα κλείσω με τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Οι μη στρατιωτικές, οι αποστολές ΕΠΑ που, είναι, που δεν είναι στρατιωτικές ξεκίνησε πραγματικότητα πριν από 6 χρόνια όταν ξεκίνησε η πρώτη μεγάλη ε, αποστολή διαχείρισης κρίσεω στη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Η EUPN, EU Police Mission, Ένωσης και ΟΗΕ. Έκτοτε αυξήθηκαν σημαντικά οι δραστηριότητε αυτές. Συνολικά έχουμε, 15, έχουμε ξεκινήσει 15 τέτοιες αποστολές. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει Δέκα αποστολές, μία από τι οποίε ε, τι διαχειρίζεται η Επιτροπή στη Μολδόβα και 9 που τι διαχειρίζεται η ΕΠΑ σε τρει υπήρου, Σε τρει δηλαδή τελείω ε, διαφορετικέ ε, σε τελείως διαφορετικές γεωγραφικές και πολιτικές συνθήκες με 2.500 άτομα προσωπικού σε όλες αυτές, συμπεριλαμβανομένου και του τοπικού προσωπικού, είμαστε πάνω από 4.000 άτομα. Οι 2.500 είναι διεθνές προσωπικό από το, τα κράτη-μέλη και από το τα κράτη που μετέχουν στην αποστολή, στις αποστολές αυτές. Όλες οι αποστολές μας βασίζονται, στηρίζονται μάλλον σε προσκλήσεις από τις υπεύθυνε αρχές, τους υπεύθυνους οργανισμούς. Ελπίζω ότι λάβατε ένα fact sheet για τις διάφορες αποστολές, ούτως ώστε να έχετε μία εικόνα των αποστολών. Οι αποστολές μας έγιναν σύνθετες όλο και περισσότερο και διαφοροποιημένες. Έχουμε τελείως διαφορετικές συνθήκες. Έχουμε αποστολή στο Αφγανιστάν, στο Κωσυφοπέδιο και τη Γεωργία. Επίσης έχουμε εμπλοκή αστυνομικών αποστολών σε δραστηριότητες του τομέα μεταρρύθμισης της ασφάλειας, μεταρρύθμισης της αστυνομίας, και μεταρρύθμιση του, του σοφρονιστικού συστήματος και του δικαστικού συστήματος, καλύπτοντας όλους τους τομείς από την ασφάλεια στην δικαιοσύνη, όλη την αλυσίδα δηλαδή της ε, πολιτικής καταστολής και εφαρμογής του νόμου. Γιατί αν θες να αντιμετωπίσεις σωστά το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίσει όλη την αλυσίδα. Οι δραστηριότητε περιλαμβάνουν απλές συμβουλευτικές δραστηριότητε, παρακολούθηση και χειρίες όπως ε, ή παρακολούθηση και χειρίες μέσα στη Γεωργία. Σε κάποιες περιπτώσεις όπως ε, κατεξαίρεση στο Κοσμοπέδιο κάνουμε και εκτελεστικές αρμοδιότητες αστυνομίας ή δικαστηρίων σε τομείς όπου οι τοπικές αρχές δεν μπορούν να έχουν εντολή να κάνουν κάτι τέτοιο. Η δύναμή μας είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους ε, επαγγελματικούς και χειριες μεσα στην γεωργια σε καποιες περιπτωσεις οπως εξαιρεση στο κοσμοπεδιο κανουμε και εκτελεστικες αρμοδιοτητες αστυνομιας πόρους από 27 κρατημέλη. Αστυνομικούς, εισαγγελείς, δικαστικούς που δουλεύουν με ενιαία προσέγγιση. Αυτό με κάνει πραγματικά περήφανο όταν διαπιστώνω ότι τι μπορούμε να πετύχουμε με τη συνεισφορά και την πολιτική βούληση των 27 κρατών μελών. Σε αυτό το πλαίσιο αυξημένο ρυθμό αποστολών και ιδιαίτερης ε, περιπλοκότητας, τα κράτη-μέλη το 2007 αποφάσισαν να δώσουν σαφή δομή ιεραρχικής ε, ε, ε, στην στις, στις μη στρατιωτικές αποστολές της ΕΠΑ. Διότι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει με, μια σύνδεση μεταξύ της πολιτικής επιτροπής που δίνει στρατηγική κατεύθυνση και έλεγχο και των αποστολών. Δηλαδή για να μπορούν να μεταφέρουν οι αποστολές τις εντολές σε πραγματικότητα. Η δουλειά μου είναι ακριβώς να σχεδιάζω, να ξεκινώ και να διευθύνω τις εννέα αυτές μη στρατιωτικέ αποστολές της ΕΠΑ ε, και λογοδοτώ στον είπα το εκπρόσωπο και στην Επιτροπή Πολιτικής και στην Πολιτική Στρατιωτική Επιτροπή απευθείας. Τα αρχικά που είπατε πρόεδρε είναι το CPCC που είναι σχεδιασμός και διεξαγωγή μη στρατιωτικών επιχειρήσεων έχουμε προσωπικό που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, αστυνομικοί, διπλωμάτες, δικαστικοί και τεχνικοί. Ένα μείγμα δηλαδή που από κοινού ε, συνιστούν μια πραγματικά θαραλέα και ε, ζωτική ομάδα. Οι αποστολές μας έχουν σαφή στόχο να σταθεροποιούμε τις περιοχές κρίσεων βελτιώνοντας την μη στρατιωτική ασφάλεια, ιδιαίτερα τις διοκτικές αρχές. Αυτή είναι η βασική μας δουλειά. Πιστεύω ότι το έργο αυτό σταθεροποίησης και παροχής μη στρατιωτικής ασφάλειας είναι προς το συμφέρον και της δικής μας ασφάλειας, της ασφάλειας ε, των πολιτών της Ένωσης. Ελπίζοντας, μάλλον θέλοντας να δημιουργήσουμε σταθερότητα και να, και να εφαρμόσουμε το κράτος δικαίου, θέλουμε να μειωθεί ο κίνδυνος να εξαχθούν οι συνέπειες των αποτυχημένων κρατών στη δική μας ε, επικράτεια. Άρα πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο αλλά ταυτόχρονα ουσιαστικό ρόλο. Ο στρατηγικός ρόλος της Ένωσης στην σταθερότητα και την μη στρατιωτική ασφαλεία έγινε κατανοητός. Ε, τρίτες χώρες μετέχουν στις, στις δραστηριότητές μας. Μεταξύ αυτών είναι σύμμαχοι. ΗΠΑ, Καναδάς, αλλά και υποψήφιες χώρες. Το γεγονός ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι διατεθειμένες να εργαστούν υπό τη δική μας εντολή είναι σημαντικό. Αυτό συνέβη στο Κωσυφοπέδιο, για παράδειγμα, που δουλέψαμε και για τα καλά. Σε αυτόν τον κατακαιρματισμένο κόσμο, όπου υπάρχουν πολλοί παράγοντες ε, και συγκρόμενες, συγκρόμενοι στόχοι πρέπει να παίξουμε έναν σημαντικό ρόλο. Αυτό είναι μια σημαντική αποστολή και γι' αυτό χρειαζόμαστε μέσα δράσεις που θα υποστηρίζουν τις διπλωματικές και οικονομικές ευρωπαϊκές προσπάθειες. Για να σας, μια, να σας δώσω μια εικόνα. Η Ευρώπη κάθε χρόνο δαπανά 11 δις στις εξωτερικές σχέσεις του πρώτου πυλώνα. Πέραν αυτών υπάρχουν και οι διμερεί σχέσει κρατών μελών που, είναι, που ανεβάζουν ακόμη περισσότερο το τελικό νούμερο. Για να έχετε μία εικόνα του μέτρου για διαχείριση κρίσεων του δεύτερου πυλώνα δαπανούμε 250 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οι αποστολές μας λοιπόν έχουν σχετικά μικρό προπολογισμό σε σχέση με τις συνολικότερες εξωτερικές δράσεις της Ένωσης. Βεβαίω, μα ικανοποιεί το αυτό και είμαστε ευγνώμονε, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερο. Τώρα, το θέμα του προπολογισμού και πά είναι καθοριστικό για μας. Μίλησα για τους 4.000 ανθρώπους που αποτελούν το προσωπικό μας και για τους οποίους είμαστε υπεύθυνοι. Για να πάρουμε κόσμο πρέπει να τους προσφέρουμε κίνητρα. Συχνά οι άνθρωποι αυτοί ζουν μακριά από την οικογένειά τους σε επικίνδυνες περιοχέ για μεγάλο χρονικό διάστημα και για χρόνου. για χρόνο κάποιες φορές. Όπως έδειξε και το EULEX στο Κόσοβο, έχουμε, όπου είχαμε την πρώτη εκτελεστική μας αποστολή, χρειαζόμαστε και εξειδικευμένο υλικό. Άρα και η υποδομή που επίση χρηματοδοτείται από την ΚΕΠΑ είναι ένα σημαντικό κονδύλι σας είπα ότι ο προπολογισμό αυτός ε, καλύπτεται, αλλά πάντα κρατάμε ένα περιθώριο για να μπορεί να αντιδράσει γρήγορα η Ένωση σε περίπτωση ανάκυψης νέας ε, κρίσης. Και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα ε, υποστηρίζει αν χρειαστούν τέτοιες νέες αποστολές. Δεν σας κρύβω βέβαια ότι υπάρχουν και προβλήματα. Ένα από αυτά αφορά τους, τους, τον χρηματοοικονομικό κανονισμό μαζί με την Επιτροπή εξετάζουμε τους κανόνες χρηματοδοτικής ε, τους κανόνες για να δούμε αν μπορέσουμε να τους προσαρμόσουμε ούτως ώστε να είναι συμβαστοί με, τους, με τις ανάγκες ε, ανάπτυξης δυνάμεων που έχουμε. Φερρυπίν, ε, αποτελεσματικά, αποτελεσματικές συμβάσεις πλαίσιο ή την αποθήκευση ειδικού υλικού γιατί ξέρετε ότι διαδικα... αν ακολουθήσουμε τις διαδικασίες ε, ανάθεσης διαγωνισμών ε, που επιβάλλει η Ένωση μπορεί να χρειαστούν 6 με 8 μήνες για να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία. Του χρόνου ο οικονομικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναθεωρηθεί. Αυτό είναι ε, μια σημαντική στιγμή για μας γιατί με τον υφιστάμενο χρηματοοικονομικό κανονισμό και τις διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών είναι πολύ δύσκολα να μπορέσουμε να συνταγιάξουμε καταστάσεις ε, όπου χρειάζεται ταχεία αντίδραση. Ελπίζω ότι αυτή η διάσταση μεταξύ πολιτικών προσδοκιών και κανονισμών, διαγωνισμών και γενικότερα οικονομικού κανονισμού θα ε, μειωθεί. Να αναφερθώ τώρα στις τρεις σημαντικότερες αποστολές που έχουμε. Δεν σημαίνει ότι άλλες δεν είναι σημαντικές, αλλά αυτές είναι οι πιο δύσκολες. Το Αφγανιστάν, πρώτα-πρώτα. Δεν θα μιλήσω επί μακρόν για την κατάσταση εκεί. Πρόκειται για ένα δύσκολο περιβάλλον. Επιπρόθεσετα, είναι δύσκολο για τρεις ακόμα λόγους. Αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά την ποιότητα της έκβασης της προεδρικής εκλογής και τη συνέπειες των εκλογών αυτών στη σταθερότητα της χώρας και άρα και της αυγανικής διοίκησης. Μετά έχουμε μια υποβάθμιση της ασφάλειας στην Καμπούλ και στην υπόλοιπη χώρα, κάτι που δυσχεραίνει την λειτουργία μας. Και τρίτον, υπάρχουν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιφέρεια. Παρά τις προκλήσεις, η αποστολή της UPOL στο Αφγανιστάν έχει βελτιώσει την επίδοσή της μετά από το δύσκολο ξεκίνημα πριν από δύο χρόνια σε κάθε επίπεδο και στρατηγικά και στη μεταρρύθμιση της αστυνομίας και σε πιο τακτικό επίπεδο. Φερρυπίν βοηθά την αναβάθμιση της αστυνομίας της Καμπούλ για να μπορέσει η αστυνομία της Καμπούλ να παράσχει καλύτερη ασφάλεια και να αντιδρά σε επεισόδια στην πόλη. Εξετάζουμε ενδεχόμενα, το ενδεχόμενο να επαναλάβουμε την ίδια, το ίδιο σχέδιο σε άλλες πόλεις του Αφγανιστάν. Επίσης, η αποστολή μας προετοίμασε την αστυνομία για την, για την υποστήριξη των εκλογών μαζί με το UNDP του ΟΗΕ. Κάτι που δείχνει ότι και ο ΙΕ μας ε, εμπιστεύεται ως εκτελεστικό, εκτελεστική υπηρεσία του και μας χορηγεί και κονδύλια. Επίσης, ε, εφαρμόζουμε το πρόγραμμα κατά της διαφθοράς στην αστυνομία και στην ε, αντικατασκοπία. Η UPOL τώρα αντι, ε, θεωρείται ως βασικός, βασική παράμετρο στη μεταρρύθμιση της αστυνομίας με ειδική εμπειρογνωμοσύνη στην ε, μη στρατιωτική διάσταση και σε, με, με σημαντικές επιπτώσεις σε όλη τη χώρα. Η Europol όμως δεν εργάζεται σε όλη την χώρα και σε διάφορες περιοχές όπου μπορεί να δραστηριοποιούνται τα λιμπάν, γιατί αυτό, αυτό κάτι τέτοιο θα απαιτούσε πολύ σημαντικότερο αριθμό και υποδομή. Ε, Δίνουμε έμφαση λοιπόν μόνο στην ε, αστυνομική και δικαστική δραστηριότητα. Η Γιούπολ αύξησε το δυναμικό της από πέρσι, 270 Διεθνής, ε, διεθνές προσωπικό και 130 ε, τοπικό, κοντά στους 400 είμαστε συνολικά. Συνεχίζουμε με τη βοήθεια της παιδείας την δραστηριότητα και συνεχίζουμε ελπίζοντας και στην δική σας υποστήριξη συχνά μας ρωτούν τι γίνεται με το συντονισμό. Το θέμα αυτό τώρα και με τη νέα αποστολή κατάρτισης του ΝΑΤΟ, το ζήτημα αυτό παραμένει βασική προϋπόθεση για να υπάρξει μια αποτελεσματική αναβάθμιση των δυνατονίτων παροχής ασφάλειας της αφγανικής αστυνομίας η νέα υποδομή ε, συντονισμού των, ε, της αστυνομία ε, στο Αφγανιστάν έχει παίξει κεντρικό ρόλο και ελπίζουμε να συνεχίσει να το κάνει. Συνολικά, στο Αφγανιστάν πηγαίνουμε προς σωστή κατεύθυνση, χρειαζόμαστε όμως περισσότερο, περισσότερους πόρους. Κόσοβο τώρα, στη Γιούλεξ. Η μεγαλύτερη αποστολή, μεγαλύτερη από όλες τις άλλες αποστολές μαζί. 1650 άτομα διεθνές προσωπικό έχουμε. Και είναι η μόνη αποστολή με εκτελεστική εντολή. Περιλαμβάνει αστυνομικούς, δικαστικούς, τελωνιακούς και ε, σοφρονιστικές υπηρεσίε. Τρεις βασικούς στόχους περιλαμβάνει και αν θέλετε να μπω σε λεπτομέρειες ε, περισσότερο σε λεπτομέρειε στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αλλά να σα πω ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι τώρα. Σταθερότητα, μεταρρύθμιση του κράτου δικαίου, και αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Τμήμα μιας ευρύτερης προσπάθειας της Ένωσης να προετοιμάσει τα Δυτικά Βαλκάνια εν ώψη μιας ε, πιθανής ένταξής του στην Ένωση. Οι τρεις αυτοί στόχοι απαιτούν ε, συνεχιζόμενες, συνεχιζόμενες προσπάθειες από τις αρχές, αλλά και από τους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η, αποστολή, η επιτυχία τη αποστολή Και χαίρο που το πολιτικό επίπεδο εμπλέκεται και αυτό ουσιαστικά. Βέβαια και το Βελιγράδι έχει ακόμα επί, επιρροή στην σερβική κοινότητα του Κωσυφοπεδίου, στο βόρειο τμήμα της ε, χώρας και ο ρόλος κατά συνέπεια του Βελιγραδίου, ιδιαίτερα και του Προεδρού είναι πολύ σημαντικός ακόμα δεν έχω και πολύ χρόνο γι' αυτό, να μιλήσω για τη Γεωργία, την πιο πρόσφατη αποστολή μας. Σε χρόνο ρεκόρ την στείλαμε, μέσα σε τρεις εβδομάδες του περασμένου Σεπτέμβρη. Η αποστολή αυτή συνέβαλε στην σταθερότητα της περιοχής. Μάλιστα ο ρωσικός στρατός αποσύρθηκε πίσω από την ε, διαχωριστική διοικητική γραμμή και έκτοτε η αποστολή μα έγινε παράγοντα σταθερότητα, κάτι που αναγνωρίζει όλο ένα και περισσότερο και η κυβέρνηση τη Γεωργία. Το πρόβλημα βέβαια παραμένει. Η αποστολή μα δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Πιστεύω ωστόσο ότι η αποστολή είναι σημαντική, κυρίως γιατί και άλλες αποστολές παρακολούθηση ε, διεθνής όπω του ΙΕ και του ΑΣΕ αποσύρθηκαν. Οπότε εμείς είμαστε οι μόνοι που είναι επί τόπου παρόντες και άρα έχουμε μια αυξημένη ευθύνη. Αποστολή μας τώρα είναι να δημιουργήσουμε μέτρα εμπιστοσύνη μεταξύ των πλευρών, κάτι δύσκολο, και να εξασφαλίσουμε ότι η Συμφωνία της Γενέβης για την, το μηχανισμό ανταπόκρισης ε, στα, στα πιθανά επεισόδια θα εφαρμόζεται. Κάτι σημαντικό επίσης στην αποστολή εκεί είναι το γεγονός ότι συνεχίζουμε τις διαδικασίες ε, διαδικασίες περιπολίες σε, σε 24 ώρη βάση και έχουμε συνάψει ειδική συμφωνία με την παροχή για την παροχή πληροφοριών από τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις. Να σας πω εντάχει και για τις άλλες αποστολές, έτσι για να έχετε μια εικόνα. Δύο αποστολές στα Παλαιστινιακά εδάφη. Μία αποστολή στο, στη μεθόδιο με, της Γάζας, μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας, η αποστολή αυτή ε, έπρεπε να αναπτυχθεί στην ράφα, αλλά έχει παγώσει η αποστολή αυτή λόγω πολιτικών προβλημάτων. Να αναφέρω τον πρόσφατο πόλεμο και τις, ε, ε, την αντιπαράθεση μεταξύ από τη μία μεριά Χαμάς Ισραήλ και από την άλλη μεριά Χαμάς Αιγύπτου, για να καταλάβετε το πρόβλημα. Έχουμε στα, έχουμε μείνει εκεί όμως, σε περίπτωση, ούτως ώστε σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία και για να ε, καθησυχάσουμε τους ε, Παλαιστινίους δεν, δεν έχουμε φύγει, δεν, έχουμε δεν θέλουμε να παγώσει η κατάσταση. Μόλις ανοίξει το, το μεθοδιακό φυλάκιο θα λειτουργήσουμε. Το άλλο λέγεται COPS. Είναι ενίσχυση της αστυνομία ε, στα Παλαιστινιακά εδάφη. Παρέχουμε ε, εμπειρογνωμοσύνη αστυνομικού και δικαστικού χαρακτήρα στην ε, δημιουργία και την ενίσχυση της ε, αστυνομίας της Παλαιστίνης. Είναι μια πολύ επιτυχής αποστολή, κάτι που αναγνώρισαν και οι Ισραηλοί και οι Παλαιστίνοι. Παρέχουμε ασφάλεια στους πολίτες στη Δυτική Όχθη και πιστεύουμε ότι η αποστολή αυτή έχει μέλλον. Έχουμε επίσης μία αποστολή στο Ιράκ, το You Just Lex, κατάρτιση 2.700 αστυνομικών και δικαστικών ε, αξιωματούχων ε, υπαλλήλων από το Ιράκ στα κράτη με, σε δομές κατάρτισης στα κράτη-μέλη. Η αποστολή δηλαδή γίνεται, κυρί, γίνεται κυρίως με έδρα της Βρυκλές και μια, ε, αντέ, μια υποέδρα στο Ιράκ, εξασφαλίζοντας ωστόσο ότι όσοι δέχονται κατάρτιση στις χώρες μας έχουν κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες που έχουν επιτόπου. Η παλιότερη αποστολή μας είναι η αστυνομική αποστολή στη Βοσνία. Έχει προταθεί η παράταση της για άλλα δύο χρόνια και ασχολείται κυρίως με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ένα θέμα που εξετάζουν και οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. Μια και η περιοχή εκεί είναι ε, φωλιά οργανωμένου εγκλήματος. Έχουμε δύο αποστολές στην Αφρική. Μία στο Κονγκό. Βοηθάμε την κυβέρνηση της, ε, του Κονγκό, Κονγκό Ζαΐ δηλαδή στην κατάρτιση της αστυνομία και έχουμε και μία πρόταση μεταρρύθμισης της αστυνομίας. Περιμένουμε να εγκριθεί το, ε, η πρότασή μας αυτή στη Γουινέα Μπισάου από την νέα κυβέρνηση. Ξέρετε ότι υπάρχει κάποιο ε, υπάρχουν μια σειρά προβλημάτων με την καινούργια κυβέρνηση, έγιναν εκλογές, ε, ε, δεν έχει, δεν έχει σχηματιστεί ακόμα η κυβέρνηση. Ελπίζουμε ότι όταν σχηματιστεί η κυβέρνηση η πρόταση θα περάσει από το Κοινοβούλιο και θα εγκριθεί. Αυτές είναι οι βασικές αποστολές. Να τελειώσω πρόεδρε τονίζοντας τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Πέντε θεωρώ. Πρώτον, ο χρόνος. Ο χρόνος είναι σημαντικός. Έχει σημασία όταν θέλουμε να φτιάξουμε την αστυνομία στα κράτη, είτε στα αποτυχημένα, είτε στα υποδιάλυση κράτη. Γιατί, γιατί πρέπει να έχουμε μία προσπάθεια που θα συνεχίζεται με, τον, με ενιαίο τρόπο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ζητούμε λοιπόν από την πολιτική ηγεσία να μας δώσει το χρόνο που χρειάζεται για να έχουμε αντίκτυπο. Δεύτερο θέμα, η αύξηση του αριθμού και του μεγέθους των αποστολών. Αυτό δεν είναι μόνο μια πρόκληση διαχείρισης για μας, αλλά και μια πρόκληση για τα κράτη-μέλη, που πρέπει να βρουν προσωπικό για τις αποστολές που αποφασίζουν. Για να σας δώσω μία εικόνα. Τα τελευταία έξι χρόνια δεκαπλασιάστηκε ο αριθμός των αξιωματούχων, που, των υπαλλήλων που χρησιμοποιήσαμε στις αποστολές μας. Χρειαζόμαστε αστυνομικούς, δικαστικούς, τελωνιακούς υψηλής ποιότητας. Χρειαζόμαστε ειδικού σε υποδομές, ειδικού σε διαγωνισμούς. Όλοι αυτοί οι ειδικοί, όχι μόνο είναι σπάνιοι, αλλά τους χρειάζονται και οι χώρες τους. μην ξεχνάτε, όταν παίρνουμε έναν αστυνομικό από το Παρίσι, μειώνεται ένας αστυνομικό, κατά ένα αστυνομικό η αστυνόμευση του Παρισιού. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα και κατά συνέπεια, αν υπάρξει πολιτική απόφαση ενίσχυσης των αποστολών μας, θα πρέπει να υπάρξουν εθνικές ρυθμίσεις για να υποστηριχθεί η αύξηση της ζήτησης προσωπικού, προσωπικού που θα έχει καταρτιστεί που θα είναι έτοιμο να φύγει αν του ζητηθεί, σε πολλές χώρες αυτές οι ρυθμίσεις δεν έχουν υλοποιηθεί. Μπορείτε λοιπόν και εσείς να μας βοηθήσετε όταν μιλήσετε με τους ομόλογους σας στα Εθνικά Κοινοβούλια, τονίζοντας τη σημασία των προκλήσεων αυτών. Τρίτη πρόκληση. Επιχειρησιακός προγραμματισμός και σχεδιασμός. Όπως ξέρετε, ο σχεδιασμός, η διαδικασία σχεδιασμού έχει αυξηθεί. Ε, η κρίση στη Γεωργία πέρσι, παραδείγματο χάρη, έδειξε ότι χρειάζεται ταχυτάτη αντίδραση για να υπάρξει επαγγελματική ταχεία αντίδραση χρειάζεται να έχουμε και συνεργάτες ε, που θα πάνε αλλά και ε, οργανωτές του σχεδιασμού της δραστηριότητας στην οποία θα πάμε. Τέταρτον, η πρόκληση των ε, διαδικασιών Ανάθεση διαγωνισμών. Όπως ξέρετε, όπω σα το είπα και νωρίτερα, οι διαδικασίε τρώνε χρόνο. Δεν μπορούμε να καλύψουμε την ταχεία προσδοκία για ανάληψη δράση. Για χρόνια ήταν ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Πέμπτη πρόκληση αυτονόητη ίσως, αλλά που καλό είναι να το τονίζω, είναι ότι οι αποστολές μας δεν πρέπει να υποκαθιστούν την διαμόρφωση πολιτικής, ιδιαίτερα εξωτερικής πολιτικής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι στέλνουμε μια, μια αποστολή και έτσι δεν λειτουργούμε διπλωματικά ή από την οπτική γωνία της εξωτερικής πολιτικής. Το αντίθετο, η εξωτερική πολιτική χρειάζεται να στηρίζει τις δικές μας αποστολές. Και αυτό είναι και η τελευταία μου παρατήρηση. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ανάπτυξη τοπικής υποδομής και τοπικής δυνατότητας υποκατάστασής μας. Πολλά εξαρτώνται από την πολιτική βούληση, την επιθυμία και την ικανότητα της τοπικής πολιτικής ηγεσίας. Αλλά αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη σε κάθε βήμα μας. Να μπορούμε να πείσουμε τους εταίρους μας να δημιουργήσουν έναν ε, τομέα ασφάλειας στη χώρα τους που θα έχει διάρκεια. Εμείς δεν μπορούμε να το πετύχουμε μόνοι μας, γιατί εμείς είμαστε στην ουσία επιχειρησιακοί παράγοντες. Χρειαζόμαστε την πολιτική βούληση των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για να πετύχουμε το στόχο αυτό. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ήταν μια πλήρης επισκόπηση και με τους συναδέλφους θα ασχοληθούμε και με διαρθρωτικά ερωθήματα και σχετικά με ορισμένες αποστολές. Θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ στις τρίτες χώρες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις διότι όπως είπατε στο τέλος το θελκτικό της ε, οργανώσεως αυτής είναι πού αναπτύσσεται και ε, πώς αναπτύσσεται ε, και οι τρίτες χώρες που συμμετέχουν σε αυτές τις αποστολές είναι μία ένδειξη της αξιοπιστίας τις οποίες χαίρουν αυτές οι αποστολές Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα θέλαμε λοιπόν ίσως να μας πείτε κάτι παραπάνω στο θέμα αυτό. Όσον αφορά την ΕΛΕΞ στο Κωσυφοπαίδιο, αναρωτιόμουν ε, όσον αφορά την αλυσίδα ε, διοίκησης ε, αντιλαμβάνομαι τι γίνεται με την αστυνόμευση δεν ξέρω τι γίνεται όμως με την δικαιοσύνη διότι δεν θέλουμε μόνο να καταρτήσουμε το δικαστικό σώμα αλλά να έχουμε και εφαρμογή δικαιοσύνης και όταν υπάρχουν τόσες ελλείψεις στο δικαστικό σύστημα όχι μόνο από την ανεξαρτησία από το 99 αλλά ε, και ε, νωρίτερα δεν υπήρχε αυτονομία, δεν υπάρχει ένα δημοκρατικό σύστημα στο κοσυφοπαίδιο οπότε όσον αφορά το έλλειμμα και τον εισαγγελέα που στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πόσο συνδέονται οι διοικήσει αυτές διότι έχω συναντήσει επανειλημμένο στο, Κόσοβο, στο ο, αξιωματούχους οι οποίοι αισθάνονται τελείως ανεξάρτητοι σε ποιον δηλαδή αναφέρονται και πώς κινούνται μέσα σε αυτό το σύνολο. Έχω δύο ερωτήσεις και η κυρία Λόζινγκ τώρα έχει ζητήσει το λόγο. Λόζινγκ, όντως είναι το όνομά μου. Ε, ήδη έχουμε συζητήσει και τσακωθεί για την συνεργασία μεταξύ πολιτικών και ε, στρατιωτικών διότι θεωρούμε ότι όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και το μέλλον η σχέση αυτή θα αλλάξει και γι' αυτό χαίρομαι κύριε Διευθυντά που έχετε τη δυνατότητα που έχουμε τη δυνατότητα να σας κάνουμε εστιασμένες ερωτήσεις. Μόνο σας είπατε προηγουμένως ε, στα σχόλιά σας ότι είναι πρόβλημα για να ξεχωρίσει κανείς τις πολιτικές από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και είπατε ότι δεν πρέπει κανείς να θεωρήσει ότι η πολιτική είναι περιττή. Στο Αφγανιστάν η σχέση των πολιτικών με των στρατιωτικών προγραμμάτων έχει κατακριθεί πολύ και γι' αυτό ρωτάω το Δεκέμβριο Δεκέμβριο 2008 υπήρξε η απόφαση του Συμβουλίου για τη Γενική Διεύθυνση 8 το στρατιω... τη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων και η διαχείριση ε, νέα πολιτική διαχείριση δηλαδή να συγχωνευθούν σε μια γενική διεύθυνση που θα καλύπτει όλο τον προγραμματισμό. Ε, αλλά ε, εκεί ε, υπάρχει μια ενοποιημένη πολιτική και στρατιωτική δύναμη μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για πολιτικές επεμβάσεις ή έχουμε καταρχήν πάντοτε ένα στρατιωτικό στοιχείο και εδώ αναφέρομαι στο Γιούλεξ, στο Κωσυφοπέδιο διότι θα ήθελα να εξετάσουμε αυτήν την πολιτική αποστολή και τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες έχουν κάνει τέσσερις ασκήσεις ε, τελευταίως τον τελευταίο χρόνο ε, επίσης ξέρω ότι και ο όρος ε, άσκηση ε, είναι αφιλεγόμενος διότι υπήρξαν πολλές φορές αμφισβητήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω εάν οι κινήσεις αυτές γίνονται από κοινού με το ΝΑΤΟ, εάν μπορούμε να μιλήσουμε για πολιτική επέμβαση και αν υπάρχει τόσο στενή διασύνδεση πολιτικών αποστολών που μετακυλούν τον πολιτικό χαρακτήρα μέχρι ένα στρατιωτικό χαρακτήρα. Συνεχίζουμε με τις ερωτήσεις. Χαίρετε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την προσέλευσή σας κύριε Διευθύντη. Έχω τρεις ερωτήσεις να θέσω. Είπατε κι εσείς, μιλήσατε για την ποιότητα του προσωπικού που είναι πολύ σημαντικό παράγον αλλά και των προσόντων του και της εκπαίδευσης training. Ξέρω ότι έχουν ε, τεθεί ερωτήματα για αυτό το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποια ακριβώς προσόντα απαιτούνται και ποια είναι η εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων. Από ό,τι γνωρίζω, κανένας από τους συμμετέχοντες ε, δεν έχει συμμετάσχει σε επιχείρηση. Αυτό είναι παράλογο. Να σχεδιάζουν επιχειρήσεις που δεν έχουν ποτέ δει στην πράξη. Δεύτερο ερώτημα. Η δυνατότητα σχεδιασμού στον ίδιο πάντα τομέα της, των δημοσίων, της διοίκησης. Πού βρίσκεστε, πού βρίσκονται τα πράγματα. Τρίτον, είναι θλιβερό ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία γυναίκα στους υπευθύνου για τις αποστολές και επιχειρήσεις. Σε πολλές χώρες, σε επιχειρήσεις που αφορούν θέματα δικαιοσύνης, γίνεται μια προσπάθεια να εκπροσωπούνται περισσότερες γυναίκες, εδώ όχι. Αυτό νομίζω είναι ένα πρόβλημα που μειώνει την αξιοπιστία μας. Και τέλος, τέταρτον δηλαδή, χτυπάω ξύλο, αλλά αν δεν εγκριθεί η συνθήκη της Λισαβόνας, τι θα γίνει με την External Action Service. Ποια είναι τα σχέδιά σας δηλαδή. Θα υπάρξει κανένα μια ειδική μονάδα διαχείρισης κρίσεων. Ευχαριστούμε κύριος Χέρνχάουζερ. Ευχαριστώ πολύ. Η ερώτησή μου είναι μάλλον θεωρητική. Δηλαδή πάντοτε αναρωτιέμαι πόσο ε, στην F10 μπορούμε να μεταφέρουμε τις πληροφορίες προς τις αρχές της Βρυξέλλες για να μπορέσει κανείς να βασίζει ορισμένες ενέργειες και όσον αφορά τις, ε, ε, το monitoring στέλνετε στις επιτόπιες αρχές και εντός 10 ημερών 10 λεπτών και στις στις Βρυξέλλες δηλαδή ε, λαμβάνουν οι Βρυξέλλες αυτές τις πληροφορίες και ποιες άλλες αρχές τις λαμβάνουν στις Βρυξέλλες. Επίσης ε, για πολιτικές ε, αποστολές όπως είναι οι ασκήσεις monitoring υπάρχουν ενημερώσεις άμεσα από αυτές τις αποστολές monitoring. Ευχαριστώ. Θα πάρω την ερώτηση του κυρίου Κύριλοφ και μετά θα κάνουμε το δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Άκουσα πολύ προσεκτικά ό,τι είπατε κύριε. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν καλύτερα να έχουμε επικεντρωθεί σε μία ή δύο χώρες και όπως πολύ σωστά είπατε ε, Αφγανιστάν και Κωσυφοπαίδιο και εκεί να εμβαθύνουμε περισσότερο και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα σοβαρά προβλήματα διότι όντως στις Ηνωμένε Πολιτείες εδώ και αρκετούς μήνες υπάρχει μία πολύ έντονη συζήτηση για του πρακτέου στο Αφγανιστάν. Και εδώ οι ε, ε, αρχές μας, ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακροφυγώς ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Και ίσως αυτό δεν είναι τυχαίο, διότι οι Αμερικανοί έκαναν ε, κακές εμπειρίες στο Ιράκ και σκέφτονται πολύ για το πώς θα κινηθούν στο Αφγανιστάν. Ακόμη και η νέα διοίκηση ο πρόεδρος Ομπάμα ο οποίος είχε αναλάβει ορισμένε δεσμεύσεις πριν τις εκλογές σκέφτεται ε, πολύ καλά πώς θα προχωρήσει ε, διότι ίσως εδώ μιλάμε μόνο για πολιτικές αποστολές αλλά πρέπει να δούμε το σύνολο διότι νομίζω ότι έφτασε η ώρα να συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά τις ε, ε, ε, την πραγματικότητα ως έχει διότι έχοντας ε, την πείρα και τις, τις ιστορικές γνώσεις για διάφορες από αυτές τις χώρες δεν ξέρω γιατί οι Βρετανοί συνάδελφοί μας δεν είναι τόσο δραστήριοι έχουν πείρα και ένα βασικό θέμα ήταν ότι το Αφγανιστάν δεν είχε ποτέ μία κεντρική κυβέρνηση. Υπήρχε ε, ε, η, ε, η αρχή από τις κοινωνικές τάξεις. Τώρα λοιπόν η χρηματοδότηση γίνεται από τους Ταλιμπάν. Οι διοικητές των προγραμμάτων ζητούν προστασία. Άρα ένα μεγάλο μέρος της χρηματοδοτήσεως πηγαίνει προς τα εκεί αντί να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Γιατί κατά τη γνώμη μου λοιπόν βεβαίως πρέπει να εκτελέσουμε την αποστολή. Δεν μπορούμε να προσπαθήσουμε να το σκάσουμε αλλά θα πρέπει ίσως να χρησιμοποιήσουμε και περισσότερους πόρους. Πρέπει όμως να ξέρουμε πού πάμε. Ευχαριστώ. Κύριε Καμπενχάουερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ε, θα πάρω τις ερωτήσεις όπως ήρθανε. Ναι. Η πρώτη σας ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, όντως είναι πολύ σημαντικά για μας και οι τρίτες χώρες βοηθούν πολύ στις αποστολές μας. Στο τέλος Αυγούστου είχαμε 200 άτομα τα οποία στηρίζονταν από αποστολές τρίτων κρατών. Δηλαδή είναι σημαντικές ε, ε, σύνδρομες και οι πλέον ε, βασικοί συνδράμοντες είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Τουρκία και σε τρίτη θέση ο Καναδάς. Βέβαια, ό,τι κάνουμε είναι υπό τον πολιτικό έλεγχο της PSC η πίεση λοιπόν πρέπει κάθε φορά να συμφωνήσει για να συμβάλλουν τα, ε, οι τρίτες χώρες. Θα πρέπει να εξετάσει κανείς τις ε, επιπτώσεις και αν υπάρξει συμφωνία ε, και μπορεί να συμμετάσχει μία τρίτη χώρα καταρτίζεται μία συμφωνία με κανόνες που είναι ίδιοι για όλους και βάσει αυτής της αρχής ε, αποδεχόμαστε τη συμμετοχή. Γενικώ είμαστε ευνοϊκοί, όχι πάντοτε, αλλά ως επτοπλίστων διότι όχι μόνο έχουμε προσωπικό αλλά έχουμε βοήθεια η οποία μπορεί να είναι πολύ σημαντική διαφέρει από τη μία χώρα στην άλλη στο Κωσυφοπαίδιο, στο Αφγανιστάν και στο Κονγκό όπου συμμετέχουν αφρικανικές χώρες. Ε, δεν θέλω όμως ε, να επεκταθώ σε αυτό, απλώς είναι χώρες που έχουν ε, συμφέροντα στην περιοχή. Προηγουμένως αναφερθήκατε στην αλυσίδα διοίκησης και αναφερθήκατε εις το εκτελεστικό σκέλος έχουμε στις χώρες μας ε, την αρχή της ε, ανεξάρτητης δικαιοσύνης και προσπαθούμε να την εφαρμόσουμε με κάποιες δυσκολίες υπάρχει όμως συνεχής διάλογος μεταξύ του δικαστικού σκέλους της αποστολής ε, και θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τους πόρους Και τέλος η εξέταση και η εκδίκαση των υποθέσεων είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασιστεί από το δικαστικό σκέλος διότι οποιαδήποτε παρεκτροπή θα πολιτικοποιούσε τη δικαιοσύνη και δεν θέλουμε κάτι τέτοιο στις χώρες μας, κατά πόσον λοιπόν σε άλλες χώρες. Όσον αφορά τις σχέσεις στρατιωτικών και πολιτικών, η κυρία Λόζιν και ο κύριος Βάλνερ ε, αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό, πρέπει να σας πω ότι συνεργαζόμενοι δεν χάνουμε την ταυτότητά μας, την διατηρούμε. Όσον αφορά την γεωργία, μας βοήθησαν όσον αφορά την διοικητική μέρημνα τις μεταφορές στις αιστείες σειράξεων, αλλά έχουμε δικές μας αποστολές, δικές, δικά μας καθήκοντα καθήκοντα, το ίδιο έχουν και οι πολιτικοί και ε, επειδή έχω πείρα σε οργάνωση τέτοιων ε, αποστολών μπορώ να σας πω ότι μας βοηθούν στην οργάνωση μεταφορών σε διάφορους ε, τομείς και δεν χρειάζεται να υπάρχουν επικαλύψεις και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επιτυχώς αυτή τη συνεργασία. Όσον αφορά την, τα θέματα της ULEX και τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ και εδώ αναφέρεστε ε, εις ε, ε, τα συλλαλητήρια παραδείγματος χάρη. Εάν συνεργαζόμαστε με τις, την τοπική αστυνομία και αν αυτή δεν μπορεί να ελέγξει την κατάσταση και μόνο αν υπάρχει ε, συνεχής και επισταμένη χρήση ε, όπλων ε, και και χρειαστεί η αποστολή να προστατεύσει τον εαυτό της τότε καλούμε τον ΝΑΤΟ να επέμβει. Μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί κάτι τέτοιο, παρόλο που η παρουσία του ΝΑΤΟ μπορεί να βοηθήσει να αποφύγουμε μία κλιμάκωση. Και αυτό είναι πολύ βασικό. Πρέπει να δώσετε το μήνυμα ότι μπορείτε να τα βγάλετε πέρα. Και θα ήθελα εδώ να συγχαρώ ε, την, ε, ε, τους, ε, τους υπευθύνους στην Πρίστινα διότι η συνεργασία ήταν εξαιρετική και μπορέσαμε να περάσουμε επιτυχώς τις διάφορες δοκιμασίες τις οποίες υποστήκαμε. Ο καθένας όμως έχει την αποστολή του με το δικό της χαρακτήρα και τη σέβεται ανα πάσα στιγμή. Όσον αφορά την εκπαίδευση, δεν είμαι ίσως ο πιο κατάλληλος για να το συζητήσω διότι αυτό είναι ο τομέας ενός συναδέλφου αλλά ε, υπάρχουν ε, πολλοί με ενδιαφέρει να είναι ο προσωπικό καλύτερα εκπαιδευμένο αυτό βέβαια είναι δικαιοδοσία των κρατών μελών και δεν μπορεί κανείς να επέμβει σε αυτή τη δραστηριότητα αλλά υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες στα πλαίσια της ΣΕΠΟΛ ε, που είναι μια αστυνομική σχολή αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω σαν κάτι τέτοιο, όπου μπορούν να δραστηριοποιηθούν και όπου μπορεί κανείς να βοηθήσει στην κατάρτιση αστυνομικών. Μας ενδιαφέρουν λοιπόν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν περισσότερο. Λοιπόν, τι άλλο. Όσο αναφορά τις ε, υπηρεσίες δράσεως, οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται είναι πάνω από το δικό μου επίπεδο. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχουν δύο κριτήρια και το λέω ε, ίσως ε, διότι εγώ δεν είμαι ε, άμεσα εμπλεγμένος. Ελπίζουμε καταρχήν ότι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την δράση μας, πράγμα το οποίο θα μας βοηθήσει και γι' αυτό έχω κάνει έκκληση να συνδυαστούν οι πολιτικές και διπλωματικές προσπάθειες με τις οικονομικές με τα οικονομικά μέσα κατά τρόπον ώστε να είμαστε πιο ευέλικτοι σε μία κατάσταση, δηλαδή οτιδήποτε μπορεί να μας βοηθήσει να εκτελέσουμε καλύτερα τις αποστολές θα είναι χρήσιμο και είναι και θέμα λειτουργικότητος. Δηλαδή, ό,τι αποφασίζεται θα πρέπει να μπορεί να αποδώσει και να μην βασίζεται μόνο σε πολιτική και γι' αυτό μιλώ για μία λειτουργική δομή. Αυτό ήθελα να προτείνω, αλλά δεν είμαι εγώ ο υπεύθυνος γι' αυτό. Um, Όσον αφορά την πληροφόρηση Πριν, πριν αναφερθώ εις ε, αποστολές ε, το ε, κέντρο πάντοτε αξιολογεί ε, τις αποφάσεις να ξεκινήσει μια αποστολή αναλόγως του τύπου της αποστολής, του εξοπλισμού με τον οποίο θα κινηθείτε, αν έχετε ιδιωτικά αυτοκίνητα κτλ. Όλα αυτά αξιολογούνται εκ των προτέρων Επίσης ε, έχουμε και ενημερώσεις ως προς την ασφάλεια, τα μέτρα που θα χρειαστούν για να προστατεύσουμε το προσωπικό μας και βέβαια η οι ε, αποστολές μας έχουν μία καθημερινή ροή ενημέρωσης αναλόγως της κατάστασης. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι ορισμένοι μιλούν και με τις πρωτεύουσές τους διότι εφόσον οι πρωτεύουσε στέλνουν κάποιον εις ε, μία αποστολή δεν ε, είναι παράλογο να συνομιλεί με τον ομόλογό του πίσω στη χώρα του και αυτή είναι η μορφή ε, της ενημέρωσης που έχουμε και έτσι τα κράτη-μέλη ενημερώνονται για τα τεκτενόμενα για να γνωρίζουν όλες τις πτυχές και εμείς διασφαλίζουμε ότι όλα αυτά ε, καταγράφονται για να υπάρχει μία ενιαία αξιολόγηση ε, για τα προβλήματα και τις προκλήσεις. Τέλος, νομίζω ότι ο κύριος Κύριλοφ μίλησε για τη σημασία που έχει η επικέντρωση της προσοχής σε λιγότερες αλλά σημαντικότερες αποστολές. Α, το συμφωνούμε, αλλά τις αποστολές τις αποφασίζουν πολιτικές αρχές, με πολιτικά κριτήρια. Εμείς εξυπηρετούμε, είμαστε στην υπηρεσία των χωρών μελών. Αν τα περισσότερα από αυτά ενδιαφέρονται για κάποιο θέμα και ληφθεί απόφαση συνενετικά για την ανάληψη μιας ε, αποστολής, την αναλαμβάνουμε όταν ενδιαφέρονται για, ιδιαίτερα για κάποιο θέμα μας χορηγούν και περισσότερους πόρους και προσωπικό. Δεν ελέγχουμε πάντοτε εμείς απόλυτα τα θέματα που εγκρίνονται. Αλλά αντικατοπτρίζουν οι αποφάσεις αυτές πολιτικά κριτήρια. Η ισότητα των φύλων είναι σημαντικό θέμα, δεν θέλω να το ξεχάσω. Πράγματι, η εξισορρόπηση των φύλων στο προσωπικό δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Έχω μερικούς αριθμούς αλλά πράγματι δείχνουν ότι καμιά φορά η εκπροσώπηση των γυναικών είναι πολύ χαμηλή, άλλες φορές είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά το προσωπικό που χορηγούν τα κράτη-μέλη το δείχνει αυτό ιδιαίτερα, γιατί εμείς μπορούμε να ελέγξουμε το προσωπικό που προσλαμβάνουμε με συμβόλαια, αλλά όχι αυτό που μας χορηγούν τα κράτη-μέλη. Για να δω... Αυτά. Είναι κάτι που είναι δύσκολο να επηρεάσουμε εμείς. Προσπαθούμε όταν έχουμε ίσα προσόντα δύο υποψηφίων αντιθέτου φίλου να παίρνουμε να χρησιμοποιούμε και το κριτήριο της εξισορρόπησης παραδείγματος χάρη τελευταία για μια αποστολή στο Αφγανιστάν αλλά είναι όντως λιγότερες οι γυναίκες και θα θέλαμε όποτε γίνεται να υπάρξει μια βελτίωση ευχαριστούμε προσθέτω ότι η συμπατριώτης μου Σιλβί Πόνς ήταν επικεφαλής μιας αποστολής στη Γεωργία πρόσφατα. Σημειωθεί το. Υπάρχουν άλλα πέντε ερωτήματα, παρακαλώ να είστε σύντομοι για να ακουστούν και οι απαντήσεις επαρκώς. Δύο λεπτά αναερώτηση. Η κυρία Αντιπρόεδρος Νικολάη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο αφορά την αποστολή την Πολωνική την αποστολή αστυνόμευσης στην Βοσνία αλλά και στην Ερζεγοβίνη. Έχει ζητηθεί η απελευθέρωση, κάποια απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων εκεί και αξιολόγηση θα ήθελα των επιτευγμάτων επιτόπου. Άλλες αποστολές είναι βέβαια διαρκούν περισσότερο χρόνο από ό,τι άλλες Μερικές φορές αλλάζει και εντολή τους κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Τι θα γίνει λοιπόν για το Κονγκό και τη Γεωργία, διότι η Γεωργία έλαβε νέα εντολή. Διότι λάβαμε νέα εντολή για αποστολή στη Γεωργία. Ο κύριος Γαλτιέρης. Ευχαριστώ. Ήθελα την άποψή σας για το βαθμό υλοποίησης του Civilian Headland Goal 2010 ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ύπαρξη ενοποιημένων, διαθέσιμων και ενοποιημένων αστυνομικών μονάδων και μία άποψη για το κατά πόσο θα έπρεπε να στείλουμε μία αστυνομική μη στρατιωτική αποστολή ΕΠΑ στην Σομαλία. Κάτι που προφανώς συνδέεται και με την διαθεσιμότητα δυνάμεων και πόρων για μια τέτοια αποστολή. Ο κύριος Βαν Μπάρεν. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία του κύριου Χουμενχάουερα. Έχω το εξή ερώτημα. Δε μας είπε ότι το θέμα είναι κυρίως η επιλογή πολιτικών προτεραιοτήτων. Δεν είναι οι ίσες όλες οι αποστολές. Η σημαντικότερη αυτή τη στιγμή είναι η αποστολή οργάνωση της αστυνομίας στο Αφγανιστάν, όπου συμμετέχει, συμμερίζεται την θετική αξιολόγηση και το Κοινοβούλιο και η Ένωση ολόκληρη, αλλά δεν φτάσαμε ακόμα στην πλήρη εφαρμογή της. Ποιο είναι το πρόβλημα. Μπορεί κανείς πάντοτε να χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο νομικό υπόβαθρο, αλλά μήπως είναι πρόβλημα πόρων, φαντάζομαι δεν είναι θέμα γραφειοκρατικών φραγμών. Μπορείτε να μας πείτε πού, πού έγκυται ακριβώς το πρόβλημα. Μήπως θα υπάρξει και για άλλες αποστολές δηλαδή. Ευχαριστώ κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να τονίσω καταρχήν το θέμα του κοσυφοπεδίου γιατί είμαι εισηγήτρια επί του θέματος. Και την περασμένη εβδομάδα μίλησα και με τον εκπρόσωπο της Γιούλεξ και με ανησυχεί ιδιαίτερα κάτι που θέλω να μου εξηγήσετε. Οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή μεταξύ Σερβίας και Γιούλεξ ενός πρωτοκόλου αστυνόμευσης δημιούργησαν προβλήματα στο κοσυφοπέδιο Όλοι λένε ότι δεν υπήρξε καλή επικοινωνία, ότι έγιναν παρεξηγήσεις δηλαδή. Η κυβέρνηση του Κωσυφοπεδίου έλαβε κάποιο μέρος, αν και στην αρχή αρνήθηκε ότι έλαβε μέρος στις διαπραγματεύσεις αυτές, αλλά και η διαδικασία συνεννόηση με τη Γιούλεξ δεν ήταν η Νομίζω ότι στο μέλλον για διαπραγματεύσεις ας πούμε για, το τελωνιακό πρωτόκολλο, για τα τελωνιακά πρωτόκολλα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και από την Γιούλεξ γιατί αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να μειωθεί η υποστήριξη του κόσμου για τις επιχειρήσεις στο κοσυφοπέδιο. Τι φρονείτε λοιπόν και γι' αυτό. Τι διαδικασίες προβλέπετε για μεγαλύτερη διαφάνεια και από την Ιούλεξ στο μέλλον. Δεύτερο ερώτημα. Υπάρχουν οι πολιτικές αποστολές αλλά αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ότι μόλις επιτευχθεί κάποια ειρήνευση αρχίζει η διαδικασία συμφιλίωσης στις χώρες όπου έχει υπάρξει σύραξη ή κάποια άλλη, κάποιο άλλο πρόβλημα και οι πράσινοι και άλλοι εδώ και χρόνια συζητούν τη την πιθανότητα δημιουργίας ενός λεγόμενου πρασίνου δικαστηρίου ε, πρασίνου σώματος παρέμβασης. Το θεωρείτε κάτι ρεαλιστικό για να διευκολυνθούν οι διαδικασίες συμφιλίωσης. Τέλος, ίσως ενδιαφέρει αυτό και άλλους συναδέλφους, ο αριθμός του προσωπικού που ασχολείται με νομικά θέματα, γιατί μέχρι τώρα μιλήσαμε για αστυνομεύσεις, τι θα μπορούσε να γίνει για να βελτιωθεί η διοίκηση εκ μέρους σας των προγραμμάτων και για θέματα δικαστικά, ας πούμε. Ευχαριστούμε τέλος ο κύριος Γκάλλαρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι. Θα ήθελα να προσθέσω μία ερώτηση σε αυτήν που έθεσε ο συνάδελφος Βαμπάλεν, ιδίω όσον αφορά την πρόσληψη, διότι ε, υπάρχουν διαφορετικές πληροφορίες τις οποίες ε, ε, συγκεντρώνουμε όσον αφορά το πώς επανδρώνουν τα διάφορα κράτη τις πολιτικές αποστολές. Είναι δυνατόν να υπάρξει ένας προγραμματισμός. Μπορείτε να μας αναφέρεται ορισμένα θετικά αποτελέσματα, δηλαδή ποιες είναι οι χώρες οι οποίες τακτικά διαθέτουν ε, ε, περισσότερα στελέχη και το αντίθετο, name and shame, για αυτούς που δεν διαθέτουν, παραδείγματο χάρη. Επίσης ε, αναφερθήκατε στους ευρωπαϊκούς κανόνες των δημοσίων προμηθειών, procurement διότι θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχει ένας πανευρωπαϊκός, μια πανευρωπαϊκή προκήρυξη διαγωνισμού και αν μπορείτε να μας περιγράψετε μια πρόσφατη περίπτωση η οποία θα εξηγήσει αυτή τη διαδικασία ε, και ίσως θα έπρεπε να συζητήσουμε με την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού του Κοινοβουλίου που είναι πολύ αυστηρή όσον αφορά τους δημόσιους διαγωνισμούς ε, επίσης αντιλαμβάνουμε ότι θα υπάρξει ένα, μια νέα γενική διεύθυνση για διαχείριση κρίσεων αλλά εκεί σταμάτησε η πρόοδος ότι κόλλησε ε, τον καθορισμό ενός διευθυντή. Μπορείτε να μας ενημερώσετε πού βρίσκεται και πότε θα ξαναξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Πρώτα η Βοσνία. Ερώτημα της κυρίας Νικολάη. Εμείς επικεντρώνουμε την προσοχή μας στο οργανωμένο έγκλημα εκεί. Η αποστολή είχε κυρίως πολιτικό, πολιτικά προβλήματα. Και νομίζουμε ότι πρέπει να προσέξουμε περισσότερο την αποτελεσματικότητά της. Δεν θα μιλήσω για την απελευθέρωση μη των θεωρήσεων, αλλά για το οργανωμένο έγκλημα μπορώ να πω ότι έχει γίνει μεν κάποια πρόοδος στην καταπολέμηση του εγκλήματος, αλλά οι υπεύθυνε αρχές για την αστυνόμευση και δίωξη του εγκλήματος στην Βοσνία έχουν κάνει κάποια πρόοδο, ίσως όχι αρκετή. Θα θέλαμε τώρα να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν πιο πολύπλοκα προβλήματα. Μπορεί εκεί να υπάρξει βελτίωση, πρέπει να υπάρξει, όπως για το δουλεμπόριο, για την παραχάραξη των ευρώ, Προσέχουμε λοιπόν ιδιαίτερα το θέμα της αντιμετώπισης πολυπλόκων εγκλημάτων, σύνθετων εγκλημάτων. Ελπίζουμε η χώρα να πλησιάσει περισσότερο την Ευρώπη και έτσι ίσως έμεσα να τη βοηθήσουμε να μπορέσει να πληρεί τις συνθήκες για μια μελλοντική απελευθέρωση των θεωρήσεων που ακόμη δεν είναι δυνατή. για το μέλλον των δύο άλλων αποστολών Γεωργία και Κονγκό και για τις δύο αυτές προβλέπεται μέχρι τα μέσα του 2010 να ολοκληρωθούν αν δεν ζητηθεί συνέχεια παράταση. Δεν μπορώ όμως να πω από τώρα ποιο θα είναι το συμπέρασμα και ούτε θα το βγάλουμε μόνοι μας γιατί και στη γραμματεία του Συμβουλίου υπάρχουν υπεύθυνοι που ασχολούνται πιο συγκεκριμένα με τέτοια θέματα. Υπάρχει και η νέα διεύθυνση για την οποία μιλήσαμε, η οποία θα προσπαθεί να συνδυάζει στρατιωτικό και πολιτικό σχεδιασμό από τα πρώτα στάδια των αποστολών για τη διαχείριση των κρίσεων ας πούμε. Μέχρι τώρα βέβαια προβλέπεται να διατηρηθεί χωριστή εφαρμογή των στρατιωτικών και των μη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Για τους λεγόμενους headline goals δεν έχω να σας πω πολλά αλλά υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών και της πραγματικότητας της καθημερινής πραγματικότητας γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε και για πιο συγκεκριμένα μέτρα διάλογο ας πούμε με τα κράτη-μέλη για εξέβρεση περισσότερου και καταλληλότερου προσωπικού. οι χώρες μέλη χρηματοδοτούν και επανδρώνουν ορισμένες αποστολές. Αυτό είναι το σύστημα που ακολουθείται μέχρι τώρα. Και ο κύριος Φαμπάλεν ρώτησε ποιο είναι το πρόβλημα. αφού πρόκειται για το Αφγανιστάν, τι ρωτάτε ποιο είναι το πρόβλημα. Και το ΝΑΤΟ έχει προβλήματα για την εξέβρεση όλων εκείνων που θα εκτελέσουν τις στρατιωτικές του αποστολές στο Αφγανιστάν. Είναι κάτι πολύ επικίνδυνο και απαιτητικό. Η δική μας ε, αστυνομική αποστολή αντιμετωπίζει όντως προβλήματα και δυσκολίες εκεί. Προβλέπονται εκεί μονοετής αποστολές που είναι κάτι ιδιαίτερα βαρύ ήδη για τους ασχολούμενους με αυτό αλλά επίσης πρέπει να σας πω ότι δεν ήμασταν οι μόνοι και οι πρώτοι που προσπαθήσαμε να οργανώσουμε μια αφγανική αστυνομία. Υπήρχαν και άλλοι οργανισμοί που ακόμη βρίσκονται εκεί και δραστηριοποιούνται. Επίσης και αυτή τη αιτήση το, της διεθνούς κοινότητας. Ο ρόλος λοιπόν της δικής μας αποστολής είναι να αποτελέσει μια συμπληρωματική προσπάθεια σε εκείνες των χωρών μελών ενώ σε άλλους τόπους σε άλλα θέατρα για να το πω έτσι επιχειρήσεων ο ρόλος της Ένωσης είναι πιο κυρίαρχος από ότι εκεί στο Αφγανιστάν μπορεί να συνδυαστεί η αποστολή αυτή με άλλες μη ενωσιακές καθαρά αποστολές. Υπάρχει και η εκπαιδευτική αποστολή του ΝΑΤΟ που επικαλύπτεται πολύ με τις δικούς μας στόχους. Επικαλύπτει τις δικούς μας στόχους. Ορισμένες χώρες δηλαδή θα χρειαστεί να χορηγήσουν και περαιτέρω χωροφύλακες από όσου έχουν ήδη χορηγήσει σε εμά. Ίσως σε έξι μήνες να βελτιωθούν τα πράγματα για μας και να έχουμε περισσότερες δυνατότητες, αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Ίσως να μην πετύχουμε το στόχο των 400 όπως έχει προβλεφθεί, αλλά συνεχίζουμε την προσπάθεια. Για την κυρία Λούνατσεκ τώρα το κοσυφοπέδιο. Ε, τι να σας πω, τα ξέρετε κι εσείς. Η διαβούλευση που ζητιέται, ναι φυσικά, προσπαθούμε να ζητήσουμε συμβουλές και διαβουλεύσεις όσο δυνατόν περισσότερο όπως με το αστυνομικό πρωτόκολλο, αλλά για πολιτικούς λόγους οι προτάσεις μας απορρίφθηκαν από τις αρχές του κοσυφοπεδίου. Υπάρχουν και διαφωνίες. Όταν προσπαθεί κανείς να συνεννοηθεί με το Βελιγράδι, δεν καταλήγει στα ίδια συμπεράσματα από ότι όταν συνεννοείται με την Πρίστινα. Η διαβούλευση λοιπόν είναι καλό πράγμα, αλλά δεν μπορεί να τα λύσει όλα. Πρέπει να υπάρξει κάποιος συνδυασμός, συμβιβασμός από όλες τις πλευρές. Που φυσικά δεν θα ικανοποιήσει πλήρως καμία. Πρέπει να έχει κανείς περιθώρια για να εφαρμόσει την κοινή λογική τουλάχιστον για την επίτευξη τέτοιων συνδυασμών. Αυτό το θέμα λοιπόν του αστυνομικού πρωτοκόλου είχε πολιτικοποιηθεί πάρα πολύ στην Πρίστινα πολύ πέραν από ότι θα ήταν λογικό γιατί για μας είναι κάτι ιδιαίτερα θετικό και θα, πρέπει να το, θα έπρεπε να το δεχτεί και η Πρίστινα αλλά θεωρήθηκε δυστυχώς σαν παραβίαση της εθνικής και πολιτικής κυριαρχίας εκεί, πράγμα το οποίο δεν είναι σωστό, δεν αληθεύει. Αυτό όμως πέρασε, είναι παρελθόν πια. Οι αρχές της Πριστίνης τώρα το δήλωσαν ρητά ότι ξεπεράστηκε πια αυτό το πρόβλημα και θα προσπαθήσουμε τώρα να κάνουμε τη δουλειά μας ε, με αξιοπρεπή τρόπο. And, um, yeah, um, για τη συμβολή των χωρών μελών που ζήτησε ο κύριος Γκάλλας δεν μπορώ ήδη εδώ από τώρα, εδώ και τώρα να αρχίσω το naming and shaming υπάρχουν ορισμένες χώρες που, που συμβάλλουν σημαντικά και τις ευχαριστώ ιδιαίτερα μερικές φορές για να το πω έτσι υπολογίζει κανείς μία η εισφορά στην προσπάθεια που είναι ανάλογη με την πληθυσμιακή σημασία της χώρας. Άλλες φορές η προσπάθεια είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι θα μπορούσε να θεωρηθεί λογικό. Ε, τι κάνουμε τότε, αρχίζουμε τις διαβουλεύσεις και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε περισσότερο ενδιαφέρον για τις χώρες χαμηλού ενδιαφέροντος. Άλλες χώρες βέβαια μας έχουν δώσει πολύ θετικά παραδείγματα, έχουν επενδύσει πάρα πολύ στις πολιτικές αποστολές, πολιτικές μη στρατιωτικές δηλαδή. Μερικές έχουν δημιουργήσει και ολόκληρη εθνική στρατηγική, άλλες όχι. Βέβαια, αν χαθούν οι θέσεις που διατίθενται για την αστυνομική δύναμη που θέλουμε να δημιουργήσουμε καταστρέφεται το πρόγραμμα ακόμη και μία θέση αν χαθεί τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα μεγάλα πρέπει να υπάρξει οικονομική αντιστάθμιση κτλ. μάλιστα τώρα για τις προμήθειες procurement δηλαδή το προηγούμενο κοινοβούλιο τα αποφάσισε αυτά και Μπορώ να σας πω δύο παραδείγματα. Ένα είναι γνωστότερο από το άλλο. Η αρχή της αποστολής μας στο Αφγανιστάν καθυστέρησε πολύ γιατί δεν είχαμε τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υλικό. Χρειάζεται συνήθως 6-8 μήνες. Αν όμως έχει ήδη φτάσει στο θέατρο των επιχειρήσεων το προσωπικό και δεν έρχονται τα υλικά, ενέρχεται το υλικό, δημιουργείται μια πολύ αρνητική εικόνα και αναξιοπρεπής. Στη Γεωργία Κάτι ανάλογο έγινε και εκεί. Και για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτής της καθυστέρησης 6-8 μηνών που απαιτείται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάστηκε να προσφύγει σε έναν μοενιαίο προμηθευτή, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε καθόλου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα θέμα ασφάλειας των προμηθειών και των αγορών μας καθώς και ασφάλεια των, της πληροφόρησης ή των πληροφοριών. Γι' αυτό νομίζω ότι και αυτοί οι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη σε, οποιαδήποτε αναθεώρηση της πολιτικής προμηθειών μας. Όχι μόνο πώς θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά και κατά πόσον υπάρχει διασφαλισμένη εκτέλεση της εντολής. Ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά για τις απαντήσεις που μας δώσετε. Ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να σας ξαναδούμε στην υποεπιτροπή μας και εύχομαι να έχετε μαζί σας και κάποιους επικεφαλής αποστολών στο μέλλον. Φαντάζομαι ότι και εμένα και τους συναδέλφους θα ενδιαφέρει να έχουμε μια απευθεία συζήτηση με τους διάφορους επικεφαλής των αποστολών στο Αφγανιστάν και αλλού. Χρήσιμο θα ήταν λοιπόν όταν ξανάρθετε να έχουμε συγκεκριμένες συζητήσεις για συγκεκριμένες αποστολές. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Συνεχίζουμε τις ε, εργασίες μας. Με χαρά καλωσορίζω σήμερα τον κύριο Τζέμι Σεϊ, Διευθυντή Πολιτικού Σχεδιασμού στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Γνωρίζει την Επιτροπή μας. Είχαμε ήδη, είχατε ήδη λάβει το λόγο πολλές φορές στην Επιτροπή αυτή, στην υποεπιτροπή αυτή στην προηγούμενη θητεία. Έχουμε στενούς και τακτικούς ε, δεσμούς με τον ΝΑΤΟ. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε την καλή αυτή συνεργασία και στο μέλλον. Πρόκειται για έναν προνομιούχο εταίρο της Ένωσης στη διαχείριση κρίσεων και η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο οργανισμών πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα για μας. Ιδίω στους τομείς που στους χώρους μάλλον όπου δούμε από κοινού ΝΑΤΟ, ε, Κωσυφοπέδιο, Αφγανιστάν κλπ ήσασταν προνομιούχος μάρτυρας των σχέσεων αυτών, αλλά και ε, παρόν στις μεγάλες εξελίξεις των τελευταίων ετών. Οπότε μπορείτε να μας διαφωτίσετε για την μεταμόρφωση της ε, συμμαχίας, τις εξελίξεις των σχέσεων της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια την αναθεώρηση της, ε, αυτού του strategic concept, της στρατηγικής ιδέας που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Θα μιλήσω στα, κόπ, στα εγγλέζικα τη μητρική μου γλώσσα. Αν ε, συμφωνείτε, γιατί πιστεύω ότι θα πω περισσότερα πράγματα σε λιγότερο χρόνο από ότι στα γαλλικά. Ευχαριστώ που με καλέσατε να έρθω σήμερα το απόγευμα. Έχετε δίκιο, δεν είναι η πρώτη φορά που είχα τη χαρά να μιλήσω στην υποεπιτροπή σας. Θυμάμαι όταν ήταν εδώ ο Καρλ Φον Βογκάου είχα τονεί πόσο δουλειά είχε κάνει για να φέρει πιο κοντά την Ένωση και τον ΝΑΤΟ και τι δυνατότητες που έδινε στο ΝΑΤΟ να μας καλεί πιο συχνά να συζητούμε τα κρίσιμα θέματα και χαίρο διότι μαζί σας ε, θα συνεχίσουμε την παράδοση αυτή. Σας ευχαριστώ οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Ένωσης, ε, δεν είναι μυστικό αυτό, είχε τα πάνω της και τα κάτω της τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτό μπορώ να πω είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την στιγμή που ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε ε, ήταν πάντα πρώτο στην δυναχορήγηση στον ΝΑΤΟ της δυνατότητα να μιλήσει και παροτρύνοντας στην ε, δημιουργία όλο ένα και στενότερων σχέσεων μεταξύ Ένωσης και ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Ελπίζω ότι Έχετε καινούργια μέλη από ό,τι βλέπω εδώ τώρα. Βλέπω και παλιούς, αλλά πολλά καινούργια πρόσωπα. Οι πόρτε μα είναι ανοιχτέ και για την επιτροπή σα και για το κάθε μέρο ξεχωριστά. Μου ζητήσατε να σα πω δύο λόγια για τη στρατηγική ε, ιδέα, αλλά πρώτα να σας τονίσω ότι θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπλακεί πραγματικά στο όλο εγχείρημα του νέου strategic concept. Ε, είναι μια στρατηγική ασφάλειας, έχετε και εσείς μια στρατηγική ασφάλεια στην Ένωση, θέλουμε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ουσιαστικά. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την όλη διαδικασία για να φέρουμε ακόμα πιο στενά, πιο κοντά τα δύο όργανα και πιστεύω ότι όπως είπε και η Μαρντλίν Ορμπλάιτ θα θέλουμε οι ειδικοί των δύο οργάνων να, κάτσουν μαζί και να διαμορφώσουν μια ενιαία προσέγγιση. Περιμένω ότι και η κυρία Ορμπλάιτ και οι ειδικοί θα έρθουν ε, μέσα Δεκεμβρίου στις Βεξελίες. Θα μιλήσω με τις υπηρεσίες σας πρόεδρε για να οργανώσουμε μια συνάντηση. Άτυπη βεβαίως, ε, αλλά που πιστεύω ότι θα είναι ενδιαφέρουσα και για τους δύο. Βλέπω, Πρόεδρε, ότι είστε πολύ θεωρητικά οργανωμένος, όχι σαν και εμένα, γιατί μου θέσετε ήδη μια σειρά ερωτημάτων για να μην ξεφύγω και για να με κρατήσετε στο θέμα σας. Στο θέμα που θέλετε να... Και θα τα ξαναπώ για να το θυμηθείτε. Πρώτον, το δόγμα του ΝΑΤΟ και την πολιτική διεύθυνση. Δεύτερον, τι γίνεται με τις αποστολές μας στο Αφγανιστάν και την αντιμετώπιση της πειρατείας στον κόλπο του Άντεν, τις στρατιωτικές ικανότητες του ΝΑΤΟ, είναι κοινέ ή συμβάλλουν κατά βάση τα κράτη-μέλη, τι γίνεται με τις σχέσεις με τη Ρωσία, ένα επίκαιρο ζήτημα προφανώς, είναι προφανές ότι η ε, λόγω και είμαι εδώ, οι σχέσεις, οι Ένωσης ΝΑΤΟ και βέβαια το strategic concept. Ξέρω ότι οι βουλευτές και να μιλήσουν θέλουν και να ακούν, οπότε θα προσπαθήσω γρήγορα να σας τα πω για να έχουμε έναν διάλογο και αν θέλετε κατόπιν να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω. Το φόγμα του ΝΑΤΟ. Δεν πιστεύω ότι οι ειδικοί που... Δεν πιστεύω ότι που θα συνειδηθούν θέλουν να ξαναδημιουργήσουν ένα νέο ΝΑΤΟ όταν του ζητήθηκε να δουν το μέλλον της οργάνωσης ή να δημιουργήσουν μια νέα οργάνωση για τον 21ο αιώνα. Προφανώ, όπως και η Ένωση και κάθε άλλος διεθνής οργανισμός, το ΝΑΤΟ μεταμορφώνεται συνεχώ τα τελευταία 20 χρόνια. Πιστεύω ότι ο τρόπος το πώς ορίζεται αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ είναι κάτι γενικά αποδεκτό από όλα τα μέλη. Τα μέλη της συμμαχίας δηλαδή δεν θέλουν να δουν ουσιαστικές αλλαγές. Το θέμα είναι πώς οι υφιστάμενες δομές θα δουλέψουν καλύτερα, πιο αποτελεσματικά και όχι πώς θα δημιουργηθεί μια νέα συμμαχία. Τι εννοώ. Πρώτον, υπάρχει μια μόνιμη συνένεση ότι η συλλογική άμυνα του άρθρου 5 παραμένει η βασική αποστολή του ΝΑΤΟ. Το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ορατή απειλή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ενεργοποίηση του άρθρου 5 για την προστασία τη επικράτεια μια χώρα αύριο, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι λιγότερο σημαντικό για τα κράτη-μέλη. Ζούμε σε ένα κόσμο όπου δεν μπορούμε πάντα να προδικάσουμε την απειλή και πολλέ φορέ ένα από αυτά που έγιναν τα τελευταία 20 χρόνια. Για τον λόγο αυτό πιστεύω ότι η όλη δουλειά της, του strategic concept ε, θα επιβεβαιώσει ότι το άρθρο 5 είναι η βασική αποστολή του ΝΑΤΟ. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να μην το βλέπουμε μόνο ως θεωρητικό αλλά και να προετοιμαζόμαστε και αμυντικά και από άποψη δυνατότητας, δυνατοτήτων να ενεργοποιήσουμε το άρθρο 5 αν ποτέ κύψει. Αν λοιπόν Ανοίγεται τώρα τη τηλεόραση και βλέπετε το ΝΑΤΟ. Είναι στο Αφγανιστάν, είναι στο Ιράν, είναι, στο Ιράκ, συγγνώμη, είναι ε, στον κόλπο του Άντεν ή στην Αφρική. Βλέπετε και την Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμπιπτόντω στον ίδιο, στους, ίδιου χώρε. χώρες. Μην πιστέψετε ότι το ΝΑΤΟ έπαυσε να είναι μια περιφερειακή οργάνωση τη Ευρώπη και ότι μετανάστευσε τρόπον την Α για να γίνει μια παγκόσμια συμμαχία. Δεν έχει τέτοιο μέλλον ούτε τέτοιε προσδοκίε στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να μπορούμε να αναλάβουμε δράση σε παγκόσμιο επίπεδο εκεί όπου το ζητά το συμφέρον των μελών μα, αλλά η ευρωατλαντική οπτική γωνία τη συμμαχία παραμένει. Βεβαίω, ε, δεύτερον, δεν βλέπω η συνένεση. Δεν βλέπω κανένα κράτος να θέλει να αποκλίνει από την αρχή της συνένεσης ε, και μάλιστα τώρα που το ΝΑΤΟ μπαίνει σε όλο και πιο επικίνδυνε αποστολέ, στο Αφγανιστάν, όπου υπάρχουν ε, θύματα πολύ περισσότερα από ό,τι σε οποιαδήποτε προηγούμενη αποστολή του ΝΑΤΟ. Η ιδέα του ότι κάθε κράτο έχει το κυρίαρχο δικαίωμα να αποφασίζει για τι αποστολέ αυτέ και δεν μπορεί να μπει στη μειοψηφία όταν είναι να στείλει στρατιώτε σε επικίνδυνε περιοχέ, γίνεται ένα, ε, μια, θεω, ένα, μια αρχή ακόμη πιο σημαντική. Η συνένεση, ξέρετε, είναι και καλή για το ΝΑΤΟ, γιατί έχουμε πολύ σοβαρέ συζητήσει. Ε, πρέπει να ε, συμφωνήσουν όλοι πριν ληφθεί μια απόφαση. Αυτό όμω σημαίνει ότι άπαξ και λαμβάνεται η απόφαση, παραμένει η συνένεση. Οι χώρε που θεωρούν ότι πρέπει να δώσουν πλήρω την άποψή του πριν συμφωνήσουν, δεν είναι τόσο πιθανό να αποσύρουν τι δυνάμει του από μια αποστολή του ΝΑΤΟ. Και το ΝΑΤΟ, παρά τι δυσκολίε όπω βλέπετε στο Αφγανιστάν, πιστεύω ότι έδειξε ισχυρή δυνατότητα παραμονή και αντοχής ε, όλων των συμμάχων. Ο Γενικός Γραμματέα στην Ουάσιγκτον προχτέ υπογράμισε ότι 23 από τις 28 χώρες υπέστησαν, είχαν θύματα στο Αφγανιστάν μέχρι σήμερα. Άρα η αρχή τη αλληλεγγύη αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Δεν μπορεί όμως να υπάρχει αλληλεγγύη χωρίς τη συνένεση. Τα δύο πράγματα πάνε πακέτο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα αλλάξει αυτό. Το τρίτο, η διεύρυνση. Το ΝΑΤΟ οι πόρτε του ΝΑΤΟ είναι ανοιχτέ πάντα. Εγώ προβλέπω ότι θα υπάρξει στο μέλλον διεύρυνση τη συμμαχία. Ήδη αναλάβαμε δεσμεύσει έναντι της Ουκρανίας, της Γεωργία, ότι θα γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ στο μέλλον. Υπάρχει ένα πρόγραμμα δράση συμμετοχή ε, που συνεχίζεται με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που είναι κοντά στην συμμετοχή με την, με την αίρεση της επίλυσης διμερών ζητημάτων. Έχουμε πολλές άλλες χώρες στα Βαλκάνια, το Μαυροβούνι και τη Βοσνία ιδίω που θέλουν να ξεκινήσουν την διαδικασία ένταξης ε, στο ΝΑΤΟ ή την ένταξη στο πρόγραμμα δάσης ένταξης, που είναι υποψήφιδα δηλαδή για μελλοντική ένταξη στο ΝΑΤΟ στην Ευρωατλαντική περιοχή, αλλά δεν μπορούν να μπουν βέβαια πριν είναι έτοιμες οι χώρες αυτές και πριν είναι το ΝΑΤΟ έτοιμο να τις δεχτεί. Βέβαια, η δυναμική της ένταξης παραμένει. παραμένει. Τώρα, για το δόγμα. Εγώ προβλέπω ότι το ΝΑΤΟ θα γίνει κυρίως μια οργάνωση της οποίας η αξία στην διεθνή κοινότητα θα είναι η δυνατότητα να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις. Δεν θα γίνουμε μια υπηρεσία μη στρατιωτικών υποθέσεων. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ε, επαναλαμβάνει το ΝΑΤΟ, αυτό που κάνει η Ένωση στην ανθρωπιστική ε, βοήθεια, στην αστυνομική συνεργασία, στην ε, δικαστική συνεργασία. Θα επανέλθω βέβαια και μετά σε αυτό, όλο. εμείς θέλουμε να έχουμε εταιρική σχέση με την Ένωση, συμβάλλοντας και συμμετέχοντας στις αποστολές αυτές, αλλά δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει πως το ΝΑΤΟ πρέπει να αποκτήσει τα στοιχεία της Ένωσης για να επικαλύψει τις δραστηριότητε. Καλύτερα είναι να παραμείνουμε σε αυτά που ξέρουμε καλύτερα. Την δυνατότητα δηλαδή χρήση στρατιωτικών δυνατοτήτων. Προφανώ θα πρέπει να γίνει με ένα διαφοροποιημένο, πιο διαφοροποιημένο τρόπο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε. Το ΝΑΤΟ τα τελευταία χρόνια κυρίε και κύριοι ασχολήθηκε με ένα τεράστιο φάσμα ε, δραστηριοτήτων ζώνες απαγόρευσης ε, πτήσεων, εμπάργο ναυτικά, ε, κατάρτιση ασφάλειας. Ε, δώσαμε την απάντηση του ΝΑΤΟ στην ανθρωπιστική βοήθεια στο Κασμί. Το 2006 είχαμε μια σημαντική αποστολή επιβολή ειρήνης στο Κοσφοβέδο και την Βοσνία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν με πολύ διαφοροποιημένο τρόπο τι στρατιωτικέ μα δυνάμει, αλλά κατά βάση ο ρόλο του ΝΑΤΟ παραμένει η ανάπτυξη των στρατιωτικών του δυνατοτήτων προ όφελο των συμμάχων και όταν μπορούμε έτσι να συμβάλλουμε ε, ουσιαστικά στην παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. Το δόγμα του ΝΑΤΟ για την ε, ε, διεύρυνση. Μέχρι, αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα. Στο δεύτερο, το, στο δεύτερο, σε τι εξετάσεις είναι, πώς πήγαμε αυτό στο πρώτο. Δεύτερον, ε, λοιπόν, δεύτερο ζήτημα, Αφγανιστάν και πειρατεία. Το Αφγανιστάν. Τώρα, ειλικρινή πρέπει να είμαστε. Προφανώ είναι μια πολύ δύσκολη και απαιτητική αποστολή. Ε, πήρε πολύ περισσότερο χρόνο από αυτό που πιστεύουμε στην αρχή όταν το 2003 έστειλε τον ΝΑΤΟ δύναμη στην Καμπούλ. Έχουμε μπροστά μα πολύ μεγάλε προκλήσει. Ε, μια ε, τοπική εξέγερση πολύ καλά οργανωμένη. Την ανάγκη να υπάρξουν παράλληλες δραστηριότητες και αλλού. Να τα βρούμε με το Πακιστάν, να σταθεροποιήσουμε την περιοχή ευρύτερα, να χρησιμοποιήσουμε ναι, ναι, ναι. τους πόρους της ΆΙΖΑΦ και τους, την ανάγκη κάλυψης των πόρων που απαιτεί, των αυξανόμενων πόρων που απαιτεί η κατάρτιση του στρατού στο Αφγανιστάν αλλά και της αστυνομία. Κυρίως δε χρειάζεται να κάνουμε πολύ περισσότερη δουλειά για να έχουμε μια συνολική σφαιρική προσέγγιση με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, εμπλεκόμενους φορείς. την Ένωση προφανώς που έχει και την αποστολή της εκεί και ασχολείται κυρίως με αστυνομική κατάρτιση ζωτικού, ζωτικής ε, σημασίας για να καλύψει το κενό ασφάλειας. Ε, αυτή τη συνεργασία και δεν είναι ε, αυτό κάτι που το λέμε συνεχώς έτσι για να το λέμε είναι κάτι που χρειάζεται για να υπάρξουν κοινοί στόχοι και να υποστηρίξουμε οι μεν τους δε στις, σε κοινέ δράσεις θα μπορούσατε να πείτε βέβαια και εσείς ότι καλό θα ήταν να είχαμε ένα ενιαίο πρόγραμμα από το 2003 όχι μόνο τώρα που έχουν μπλέξει και όλες οι στρατηγικές αναθεωρήσεις. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Η μόνη βιώσιμη στρατηγική εξόδου καρνάτου είναι η αυγανοποίηση, δηλαδή η προοδευτική χορήγηση αρμοδιοτήτων στις αυγανικές και ευθυνών στις αυγανικές αρχές. Ήδη μεταφέραμε αρμοδιότητες στους Αφγανούς στην περιοχή της Καμπούλ οι Υπουργοί Αμήνης που θα συναντηθούν σε δύο μέρες στην Πρατισλάβα θα συζητήσουν ε, τις διάφορες φάσεις ε, της μετάβασης. Ε, ούτως ώστε να υπάρχει μια βιώσιμη στρατηγική εξόδου, όχι, όχι έξοδος, στρατηγική εξόδου, μην μπερδεύετε τα δύο. Αυτό θα περάσει και από, την, και από ένα πρόγραμμα κατάρτισης, στο οποίο θα μετάσχουν όλες οι χώρες. Η έξοδος από το Αφγανιστάν απαιτεί ωστόσο περισσότερους πόρους από αυτούς που είχαμε εξοφλήσει. Επίσης, αν θέλουμε να φύγουμε πρέπει να έχουμε τους πόρους τώρα, ούτως ώστε να ολοκληρώσουμε την κατάρτιση και να βοηθήσουμε τους Αφγανούς να αυξήσουν την εσωτερική διακυβέρνηση. Δεν λέω λοιπόν ότι είναι πανάκια ε, ή ε, αυτό για να απαντήσουμε στα ζητήματα του Αφγανιστάν, αλλά είναι σημαντικό για να υπενθυμίσουμε στον κόσμο γιατί είναι σημαντική η αποστολή αυτή και τι συνέπειε θα είχε η αποχώρησή μα που θα άφηνε του Ταλιμπάν να ξαναπάρουν την εξουσία στην Καμπούλ όπω ε, το είχαν κάνει πριν το 2001. Πειρατεία. Δεν είναι ευθύνη του ΝΑΤΟ αυτή όπως το Αφγανιστάν, διότι εμπλέκονται πολλοί παράγοντες το τομέα αυτό. Η Αταλάντη, η Ευρωπαϊκή Αποστολή που πήρε παράταση ενό έτου άλλωστε, είναι αποστολή με καλύτερου πόρου από την αποστολή του ΝΑΤΟ και σε ό,τι αφορά τι πληροφορίε και σε ό,τι αφορά την αεροπορική υποστήριξη και τις νομικές ε, ρυθμίσεις με χώρες όπως την, ε, και την Κένια που προβλέπει την ε, κράτηση των πειρατών. Δεν αντικαθιστούμε την Ένωση, Θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να συμπληρώσουμε. Πιστεύω ωστόσο ότι η πειρατεία απετέλεσε ένα ενδιαφέρον παράδειγμα για το πώς μπορεί να συνεργαστεί καλύτερα το ΝΑΤΟ με την Ένωση. Γιατί για πρώτη φορά είχαμε κοινό στρατηγείο τον Όρφορ, στον στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ένας Βρετανός, ε, ήταν δίπλα-δίπλα στο δίπλα τραπέζι με τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αποστολής, επίσης Βρετανό. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Δεν πρέπει να τσακωνόμαστε για τα ίδια πλοία ή για τα ίδια στοιχεία. Αυτό που ε, ε οι διπλωμάτες μερικές φορές αποκαλούν double dipping, δηλαδή να βάζουμε και δύο το χέρι στο ίδιο ε, το ίδιο κομματάκι κρέας. Αυτό σημαίνει ότι ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες όπως έγινε πρόσφατα. Τρίτο ζήτημα. Δυνατότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρκετές, ούτε και εμείς έχουμε. Ε, είναι Ούτε εμεί έχουμε ούτε αυτοί, το είδαμε και στο Τσάτ, το είδαμε και στο Αφγανιστάν. Οι ίδιε ε, ωστόσο δυναμίε εμφανίζονται και στα ε, και σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Ε, ελικόπτερα, οι μηχανικοί, μονάδες υποδο... μηχανικές μονάδες, αεροσκάφη, ε... για τη χρηματοδότηση, προβλήματα κοινή χρηματοδότηση που μπορεί να κρατήσει ολόκληρη δομή, ολόκληρο, ολόκληρο άθροισμα μονάδων. Περικοπές στου προπολογισμού Άμυνα. Δεν μπορούμε ε, να χάνουμε, να διασπαθίζουμε τους πόρου Και το ΝΑΤΟ και η Ένωση έχουν το πρόβλημα ότι πολλέ δυνάμεις μας δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Ο Ρουντ Λούμπερ, αν το θυμάστε, γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ παλιά, έδινε στοιχεία για το πολύ μικρό ποσοστό ευρωπαϊκών δυνάμεων που έχουν εκπαίδευση και εξοπλισμό για να βγουν εκτός χώρας. Οι επενδύσεις μας εν ε, παραμένουν επενδύσεις της εποχής του ψυχρού πολέμου. Δεν βαριές υποδομές χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης ε, παρότι αυτό το είχε πει πολλά χρόνια πριν ε, ισχύει και τώρα. Και οι δύο οργανώσεις λοιπόν πρέπει να μπορέσουν να κάνουν τα εξή. Πρώτον, να εξασφαλίσουν ότι τα κράτη-μέλη όταν ε, καταρτίζουν τα εθνικά μηδικά του προγράμματα να λαμβάνουν υπόψη τι απαιτήσει τη Ένωση και του ΝΑΤΟ. Δεύτερον, να αναζητήσουν συνέργεια και να μην, επαναλαμβ... Ε, επικαλύπτουν ε, το ένα το άλλο τις ίδιες δραστηριότητε, αλλά να δουν πώ μπορεί να συμπληρώσει το ένα το άλλο. Παράδειγμα, κατάρτιση των ε, μαχητικών μονάδων της Ένωσης. Μπορεί να γίνει με, ε, ε, μονά, με κονδύλια του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν σημαίνει ότι να, δεν θα μπορούν οι, οι δύο, τα δύο όργανα να, να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα τις δυνάμεις τους, αλλά αυτό θα έχει πολύ φθηνότερο κόστος. Και χρειαζόμαστε επίσης να εξασφαλίσουμε ότι οι ικανότητες που διαθέτουμε είναι πραγματικά διαθέσιμες και, στις δύο, και στους δύο οργανισμούς. Παρότι παραμένουν κατόνομα υπό τον έλεγχο της μίας. Φερρυπίν, το ΝΑΤΟ δύο φορέ χρησιμοποίησε το Eurocall. Αυτή ήταν η επικεφαλή των επιχειρήσεών μας. Ο κύριος Ντεχόψεφτερ, ο το παλιό αφεντικό μου, είχε προτείνει να είναι έτοιμο το ΝΑΤΟ να ε, μοιραστεί με τις ευρωπαϊκές αποστολές το μεταφορικό αεροσκάφος C-17. Αρχίζουμε λοιπόν και βλέπουμε πού μπορούμε να συνεργαστούμε. Καθώς δημιουργούμε κοστοποτελεσματικές δυνατότητες. Ρωσία. Ναι, ας προχωρήσουμε. Πολλοί θα θυμηθήκατε την ομιλία του κύριου Ράσμου την περασμένη εβδομάδα. Σήμερα, το τώρα που ερχόμουν, συνεχιζόταν εκείνη τη στιγμή μια συνάντηση του ΝΑΤΟ με, την, με, τους, πρέπει να υπάρχει μια καλή σχέση ΝΑΤΟ και, ε, και Ρωσίας. Πόσο μάλλον που γιορτάζουμε σε λίγες εβδομάδες τα 20 χρόνια της πτώσης του τείχους του Βερολίνου. Πάρα πολλά όνειρά μας υλοποιήθηκαν την τελευταία 20 ετία για την επανένωση σε ειρηνικό πλαίσιο της Ευρώπης. Η Ρωσία, ωστόσο, είναι μια χώρα που δεν θεωρεί ότι είναι ικανοποιημένη από τις σχέσεις της με τον ΝΑΤΟ και ευρύτερα με την Ευρώπη. Δεν έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα ασφάλειας ε, με τη Ρωσία, έτσι τουλάχιστον όπως το αισθάνεται η ίδια. Άρα πρέπει να γίνει δουλειά. Και νομίζω ότι η 20η επέτειος ε, της πτώσης του τείχους είναι ένα καλό κίνητρο να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να φέρουμε κοντά μας στη Ρωσία. Αυτό μπορεί να γίνει για το ΝΑΤΟ, διότι η συνεργασία με το ΝΑΤΟ θα είναι πολύ χρήσιμη για να λυθούν θέματα όπως η παροχή ενέργειας, η αύξηση των όπλων, η αντιμετώπιση της δημοκρατίας. Χρειάζεται το ΝΑΤΟ την Ρωσία. Φερρυπίν στι διαπραγματεύσει για ε, ο, διόδους τράνζιτ. Ε, ε, Άρα πρέπει να συνεχιστεί. Βεβαίως αυτό δεν θα εμποδίσει το ΝΑΤΟ. Το είπε αυτό ο κύριος Ράσμουσεν ε, μιλώντας ειλικρινά στην Ρωσία. Δεν θα μας εμποδίσει να έχουμε την άποψή μας όταν διαφωνούμε. Αυτό που θέλουμε να έχουμε και δεν το πετύχαμε μέχρι τώρα με τη Ρωσία είναι να υπάρχει μια διαδικασία όπου μπορεί να υπάρχουν διαφωνίε χωρί να, μπλοκάρει, να μπλοκάρει για μήνε ολόκληρη η διαδικασία και όπου θα μπορούμε να συνεργαστούμε σε τομεί όπου θέλουμε να συνεργαστούμε και παρά τα αυτά να έχουμε διαφωνίε σε, άλλο, σε άλλα επίπεδα. Το είπε και ο Γενικός Γραμματέας. Πρέπει να εστιάσουμε τις σχέσεις μας δίνοντας έμφαση στα θετικά και όχι στα αρνητικά όπως πάντα. Για να σας πω την αλήθεια, πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε μια συμφωνία για να διασφαλίσουμε τους Ρώσους ότι αντιμετωπίζουμε τις ενσυχίες τους για μια ευρωπαϊκή ασφάλεια και ότι δεν τους αγνοούμε. Αυτό είναι η ιδέα του προγράμματος Μετβέντεφ για την Ευρωπαϊκή ε, ε, Συνθήκη Ασφάλειας πρέπει να καλύψουμε τις θεμητές ανησυχίες των Ρώσων. Ταυτόχρονα η Ρωσία θα ήταν έτοιμη να συνεργαστεί με το ΝΑΤΟ στους τομείς της πειρατείας που θεωρούμε ότι είναι αναγκαίοι. Όπως σας είπα, ο κ. Ζάσμουσεν συναντηθήθηκε με τον κ. Λαυρόφ στην ε, Νέα Υόρκη. Συμφωνήσαν σε μια σειρά θεμάτων, ε, εμπλοκή στο Αφγανιστάν, αξιολόγηση των σημείων διαφωνίας και συμφωνίας και θα δούμε πώς θα προχωρήσει το πράγμα τους επόμενους μήνες. Τώρα, σχέσεις με τη, μεταξύ ΝΑΤΟ και Ένωσης. Πόσες ώρες έχετε, θέλετε να σας τα πω Συνοπτικά ή εκτεταμένα. Συνοπτικά. Να σας τα πω, αλλά είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα. Εν ολίγης, πιστεύω ότι έχουμε μια ευκαιρία, καλή ευκαιρία, να έρθουν κοντά οι δύο θεσμοί. Όχι να συγχωνευτούν, κάθε οργανισμός έχει διαφορετική δραστηριότητα. Άλλο η Ένωση, άλλο το Η Ένωση ξεπερνάει τον τομέα της ασφάλειας, ε, αλλά είμαστε κοντά. Και γιατί είμαστε πιο κοντά. Αυτά που σας λέω είναι προσωπική άποψη, αλλά ελπίζω, και όλοι το ελπίζω φαντάζομαι, ότι η συνθήκη της Λισαβόνας θα κυρωθεί και θα υλοποιηθεί γρήγορα. Διότι όχι μόνο θα δώσετε εργαλεία στην Ένωση στον τομέα της ε, κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και έτσι θα μπορέσει ευκολότερα και να συζητήσει γραφειοκρατικά και διπλωματικά με τον ΝΑΤΟ, αλλά και γιατί πλέον θα υπάρχει ένα νέο πλαίσιο που θα λέει να η Ευρώπη από εδώ και πέρα, άρα από εδώ, με βάση αυτό θα λειτουργήσουμε. Δεύτερον, η Γαλλία, όπως όλοι γνωρίζετε, επανεντάχθηκε στο στρατιωτικό σκέλο του ΝΑΤΟ, κάτι που σημαίνει ότι σχεδόν καμία μεγάλη χώρα στην Ένωση δεν βλέπει να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ ισχυρού ΝΑΤΟ, ισχυρής Ένωσης. Ότι το ένα δηλαδή θα υπονομεύσει το άλλο ή ότι το ένα θα αποδυναμώσει το άλλο. Πρόκειται για μια ευκαιρία. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα Ένας από τους στρατιωτικούς ηγέτες του ΝΑΤΟ είναι ένας πτέραχος Γάλλος. Και άλλωστε αυτό, αυτή την άποψη έχουν πλέον και οι Αμερικανοί, όχι μόνο επί Ομπάμα και επί Μπούς. Έλεγαν ότι μια αδύναμη Ευρώπη είναι ένα αδύναμο ΝΑΤΟ. Θεωρούν η άποψη της Αμερικανικής κυβέρνησης είναι ότι η βελτίωση, η ενδυνάμωση στρατιωτικά ε, ε, στον τομέα της ασφάλειας της Ευρώπης είναι καλό για τον κόσμο. Λοιπόν, οι παλιές κουβέντες ότι το ένα θα φάει το άλλο έχουν τελειώσει. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε ότι θα μείνουμε άνεργοι στον τομέα της ασφάλειας αύριο. Και αυτό ισχύει και, τους δύο, και, τις δύο, και για τον Άτομο και για την Ένωση. Βεβαίως, προφανώς υπάρχει μία έμεση κατανομή αρμοδιοτήτων. Οι βαριές δουλειές, στρατιωτικές δουλειές, Αφγανιστάν σήμερα, Βοσνία το 1995, ανήκουν στο ΝΑΤΟ. Αντίθετα η Ένωση έχει ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων, κυρίως στους μη ε, στο μη στρατιωτικό τομέα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει έτσι, θεολογική διαίρεση μεταξύ των δύο και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσεται άρα καμία κατανομή δεν θα μείνει ως έχει για πολύ. Οι διπλωμάτες και η πολιτική ηγεσία έχουν μυαλό. Μπορούν να καταλάβουν ποιο οργανισμός είναι ο πλέον ενδεδειγμένο για να αναλάβει την ηγεσία. Ο άλλο θα πρέπει να το υποστηρίζει επικοδομητικά. Και πρέπει να σα πω ότι Πολλοί εδώ αγωνιούν ε, σε συνέδρια και σε σεμινάρια για τις σχέσεις ε, Ένωσης ΝΑΤΟ. Εγώ πιστεύω ότι η κατάσταση των πραγμάτων θα μας επιτρέψει να συνεργαστούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε ωστόσο άμεσα. Πρώτον, να αναγνωρίσουμε ότι το Βερολίνο ΣΥΝ, ζητώ συγγνώμη για, και τα καινούργια μέρα, δεν μπορώ να αποφύγω τις, ε, την ξύλινη γλώσσα. το Βερολίνο 2, το Βερολίνο ΣΥΝ λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δανείζεται τις ικανότητες του ΝΑΤΟ και κάνει τις αποστολές του ΝΑΤΟ σε άλλες περιοχές. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο ωστόσο. Όλο και πιο συχνά διαπιστώνουμε ότι βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο. Πειρατεία, ε, Κωσυφοπέδιο, Αφγανιστάν, Βοσνία. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία συμφωνία που θα λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι πρέπει να συζητούμε όταν είμαστε μαζί, έστω και να κάνουμε διαφορετικές δράσεις. Άλλο στην αστυνομία, άλλο στο στρατό. Και δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στη Βοσνία που είναι η μόνη αποστολή Βερολίνο ΣΥΝ. Και αλλού θα πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο για περιοχές στις οποίες είμαστε και οι δύο. Δεύτερον, χρειάζεται να έχουμε τακτικότερες επαφές μεταξύ του του εκπροσώπου, του κυρίου Σολάνα, και του Γενικού Γραμματεία του ΝΑΤΟ. Βεβαίως και, και συναντιόνται, αλλά πρέπει να έχουν μια πιο συστηματική προσέγγιση με κοινή ανάλυση, κοινή αμοιβαία ενημέρωση, κοινέ ε, ατζέντε, κοινή μερίσια διάταξη. Η Γαλλική Προεδρία πρότεινε ένα είδος ε, ομάδας εργασίας ε, που το ακολούθησε και η Σουηδική ε, Προεδρία. Κάτι τέτοιο πρέπει να συνεχιστεί. Τρίτον, καθώς η Ένωση αποκτά μεγαλύτερη εμπειρία σε τέτοιες δραστηριότητε. το ΝΑΤΟ θα ήθελα να ακούει από εσά περισσότερο για τα διδάγματα που δράτεται. Πρόσφατα υπήρχε μία πρόταση να ενημερώσει η Ένωση το ΝΑΤΟ για την επιχείρηση Αταλάντη. Μια τελευταία παρατηρήση, Πρόεδρε. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία στις στρατιωτικές, στις δυνατότητές μας, ούτως ώστε π.χ. αν ο ένας οργανισμός έχει ένα καλό αμυντικό πρόγραμμα, να μην ξαναπληρώνει ο άλλος οργανισμός τα ίδια για το ίδιο εργαλείο. Πρέπει να ανταλλάσσουμε περισσότερες πληροφορίες για να ενισχύσουμε τη συνεργασία. Αυτό θα θέλω να δω. Τέλος, σε αυτό το πολύ σύντομο, σε αυτή την πολύ σύντομη επισκόπηση που τους περισσότερους τουλάχιστον σας κράτησε ξύπνιους, ή το strategic concept. Δύσκολος όρος αυτή η στρατιωτική, η νέα έννοια της στρατιωτικής δράσης. Ξέρουμε ότι πρέπει να τελειώσει τέλη του έτους η συζήτηση για το θέμα. Πάντως ξέρω ότι πέντε πράγματα θα χρειαστεί να δουν οι ειδικοί. Ξέρω ότι θέλω να φτάσει στις ερωτήσεις. Πρώτον, ισορροπία μεταξύ δραστηριοτήτων του άρθρου 5 και εκτός άρθρου 5. Πώς θεωρητικά και πολιτικά μπορεί το ΝΑΤΟ να εξισορροπήσει την απέτηση άμυνας του ευρωπαϊκού εδάφους όπως λέει ο κύριος Βαν Όντεν που φαντάζομαι τον ξέρετε παλιός συνάδελφος να υπερασπιστούμε το κάστρο μέσα στο κάστρο και να πάμε έξω από το κάστρο ταυτόχρονα. Κάποιοι σύμμαχοι δίνουν έμφαση στη μία διάσταση, δηλαδή την άμυνα του εδάφους και άλλοι στην ε, δραστηριότητα εκτός Ευρώπης. Δεν είναι αντιφατικές οι δύο προσεγγίσεις, αλλά έχουν ε, διαφορετικές ε, φιλοσοφίες αν θέλετε. Ο ένας λέει ισχυρές δυνάμεις, στέρες, έτσι, σταθεροποιημένες δυνάμεις, ε, στρατηγία κλπ. Οι άλλοι λένε μονάδες ετοιμοπόλεμες ανά τον κόσμο. Επίσης, εταιρικές σχέσεις. Ό,τι και να κάνουμε τώρα το κάνουμε με εταίρους. Προφανώς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη αλλά και όλο ένα και περισσότερο χώρες του Περσικού κόλπου, της Βορειοαφρικής. Άλλες, έχουμε 20 χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, από Σιγκαπούρη και Αυστραλία. Η Σιγκαπούρη είναι και στο Αφγανιστάν. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε παγκόσμια παρέμβαση χωρίς τους εταίρους αυτούς. Διότι ό,τι και να κάνουμε απαιτεί υπερπτήσεις, διελεύσεις, προσωρινές αεροπορικές βάσεις, κουλουπού. Τώρα πώς κρατάει τις σχέσεις αυτές στο ΝΑΤΟ. Πώς αποφεύγουμε να δώσουμε την εντύπωση ότι το θεωρούμε δεδομένο. Ότι οι χώρες αυτές συμβάλλουν, είναι υποχρεωμένες να συμβάλλουν, να έχουν θύματα, αλλά να μην μετέχουν στις συζητήσεις, στις αποφάσεις. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ορισμένοι από τους μηχανισμούς που διαμορφώσαμε στη δεκαετία του 90, το Partnership for Peace ας πούμε, και που είχαν φτιαχτεί για, μια, για ένα ΝΑΤΟ ευρωκεντρικό, μπορεί να μην είναι αναγκαία, δεν να μην είναι τα ενδεδειγμένα για μια πιο παγκόσμια εικόνα του ΝΑΤΟ του 21ου αιώνα. Τρίτο θέμα. Η Μόνς. Πρότυπα. Και ένα θέμα που μέχρι τώρα δεν μας είχε απασχολήσει μας σαν το πολύ. Όσοι παρακολουθείτε ωστόσο τις συζητήσεις για την ασφάλεια, θα δείτε ότι έχει αυξηθεί τεράστια η νομοθετική προσέγγιση. Συμβάσεις για τα όπλα, δικαστήρια, πρωτοβουλίες κατά της αξάπλωσης των όπλων, όπλα μαζικής καταστροφής και προφανώς η ασφάλεια του 21ου αιώνα σημαίνει όχι μόνο να περιμένουμε να μας επιτεθούν, αλλά να διαμορφώσουμε και το πλαίσιο, να δημιουργήσουμε κανόνες, να εμπλέξουμε νέες χώρες, ε, Ινδία, Κίνα, να εξασφαλίσουμε ότι η συνθήκη μη διάδοση θα ανανεωθεί του χρόνου, ότι θα μειωθούν τα όπλα από εμά που δεν θέλουμε να έχουν και άλλοι. Και προφανώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλέκεται σε πολλούς τομείς όπως και ο ΙΕ. Και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αποφασίσει τι θέλει, να εμπλέκεται ή να αντιδρά στους τομείς αυτούς. Εμείς έχουμε μια σφαιρική στάση, πολύ καλό, αλλά κάτι τέτοιο δεν απαιτεί, δεν σημαίνει σφαιρική προσέγγιση. Το ότι θέλουμε να είμαστε πλούσιοι δεν σημαίνει ότι θα γίνουμε πλούσιοι. Δεν περιμένουμε το τζίνι να βγει από το από το λιχνάρι, πρέπει να αναλάβουμε και εμείς δράση. Και τέλος, χρειάζεται να εξετάσουμε πώς θα εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα μπορεί να παράσχει τις ικανότητες για ένα ευρύτερο φάσμα απαιτητικότερων αποστολών. Προφανώς λοιπόν τους επόμενους μήνες οι ειδικοί θα δουλέψουν πολύ εξετάζοντας όλα αυτά τα θέματα. Με άλλα λόγια, όπως όλοι μας και το ΝΑΤΟ έχει μπροστά του πολλές προκλήσεις έχει πολλές δυνατότητες. Υπάρχει ένα κενό προφανώς μεταξύ της, ε, των δυνατοτήτων και των ε, προκλήσεων και η πρόκληση για μας είναι να φέρουμε κοντά τις δύο αυτές έννοιες. Ε, ξέρω ότι μίλησα πολύ, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Ελπίζω στόσο να σας δημιούργησε αρκετά ενδιαφέροντα για να τα καλύψετε με μια σειρά ερωτήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Προφανώ θα τεθούν. Δεν με στενοχωρεί καθόλου το ότι σα είχα θέσει εκ των προτέρων ορισμένα ερωτήματα γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσε οι απαντήσει. Αλλά δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε και το χρόνο των διερμηνών και ήταν και αυτό ένα τρόπο. Λοιπόν, μου φάνηκαν πολύ ικανοποιητικά αυτά που είπατε για τις σχέσεις Ένωσης και ΝΑΤΟ Δυστυχώς δεν ήταν όλοι οι συνάδελφοι παρόντες για να τα ακούσουν γιατί συμφωνώ ότι πρέπει να μην είναι δογματική η αντιμετώπιση μας. Ιδιαίτερα αναφερθήκατε στην αλλαγή της τάσης της Γαλλίας, που με ικανοποιεί και εμένα ιδιαίτερα. Λοιπόν, σειρέ έξι ερωτήσεων. Ο κύριος Φόμποντα πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όπως ε, συνήθω είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία σας πολλά σχόλια εκ των οποίων δύο είναι τα βασικά καταρχήν να υπάρχει ε, στενή συνενδαξία και επαφή με την ομάδα η οποία καταρτίζει τη νέα στρατηγική για τον ΝΑΤΟ και ίσως ε, υπάρχουν ιδέες τις οποίες μπορούμε να περιλάβουμε σε έκθεση που αυτά είναι πολύ σημαντικά και δεύτερον η Ρωσία η ομιλία του νέου Γενικού Γραμματέα ήταν πολύ θαραλέα. Μετά πήγαμε στη Μόσχα. Ε, βέβαια δεν ήταν εύκολο για την Ρωσία. Είπαν, ε, είδατε δεν μας θέλουν, οπότε η θέση είναι σαφής. Και από το ο Ράσμουσεν, ο Ομπάμα κάνουν προσφορές, προτάσεις και πάντοτε ε, ε, δεν είναι, δεν είναι αναγκαστικά η ύπαρξη ενός προγράμματος προκαθορισμένου αλλά η επιθυμία για διάλογο και εδώ αναφέρομαι στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία και την Γεωργία ε, είναι θέματα που θα συζητηθούν με τη Ρωσία ή θεωρείτε ότι είναι θέματα που δεν πρέπει να συζητηθούν με τη Ρωσία διότι η Ρωσία αν συζητηθεί ε, και αποτελεί μέρος του διαλόγου θα πρέπει και οι ε, χώρες οι παραμεθόριες να μπορούν επίσης να συζητηθούν. Ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ. <clears throat> Ε, θα ήθελα εδώ να εστιαστώ στη σχέση μεταξύ ε, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν πρέπει να είμαστε πολύ θεωρητικοί αλλά ε, ρεαλιστές και θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα όπως το πρόγραμμα Αταλάντη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η πρώτη που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό και και κάποια στιγμή είδαμε εμπλοκή και του ΝΑΤΟ επιπλέον. Αυτό ίσως εξηγεί πώς μπορούμε να συντονιστούμε καλύτερα και να μην δίδουμε τουλάχιστον την εντύπωση ότι γίνεται εκ του παραλίλου κάποια κίνηση και ο ένας ζηλεύει για το ότι κάνει ο άλλος ή ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους γίνονται αυτά. Όσον αφορά την ε, ε, ε, στρατιωτική δύναμη του ΝΑΤΟ από τη μία μεριά ε, βλέπουμε ότι τώρα στο Αφγανιστάν υπάρχει η προσπάθεια να αναπτυχθεί και το πολιτικό σκέλος. Αυτό συνάδει με την περιγραφή ε, που έκανε στη μηνιαία συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος Ράσμουσεν ο οποίος είπε ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ νατο και ευρωπαϊκής ενώσεως εάν μπορέσουμε να συντονίσουμε την ε, στρατιωτική δύναμη και ε, την διατλαντική εμπλοκή του νατο με το πολιτικό σκέλος της ευρωπαϊκής ενώσεως. δηλαδή ε, εννοείται ότι η ευρώπη θα προσφέρει τη χρηματοδότηση και το πολιτικό σκέλος ή ε, θα προσλαμβάνει οικονομικά η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ΝΑΤΟ για να τις κάνει τις δουλειές. Ε, ίσως λοιπόν θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα και να μας το εξηγήσετε. Ευχαριστώ. Κύριος Βαμπέλ. Θα ήθελα κύριε Σύ να σας θέσω το εξής ερώτημα. Αν δείτε ποια είναι τα καθήκοντα του ΝΑΤΟ, θα καταλάβετε ότι πρόκειται για συνεργασία Καναδά, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης. Όχι μόνο για την ανάπτυξη μιας, ενός στρατηγικού σχεδίου, αλλά και ως προς τη διοικητικά. Θα έπρεπε λοιπόν να αναρωτηθούμε αν οι επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν πρέπει να θεωρηθούν σαν επιτυχία ή αποτυχία του ΝΑΤΟ. Δεν θα ήταν καλύτερο, σωστότερο να μην χρησιμοποιούμε τον ΝΑΤΟ ως οργάνωση καθεαυτήν, να χρησιμοποιούμε μόνο τις εγκαταστάσεις και τους πόρους του και να το χρησιμοποιούμε απλώς ως συντονιστικό όργανο. Γιατί η αποτυχία της αποστολής στο Αφγανιστάν μπορεί να, φτάσει, να καταστρέψει τον ΝΑΤΟ. Ίσως λοιπόν τα καθήκοντα του ΝΑΤΟ να πρέπει να είναι μάλλον συντονιστικά παρά επιχειρησιακά. Κυρία Λόιζινγκ. και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εκτενή παρουσίαση. Ε, σε κάποιο σημείο είπατε ότι η ιδέα της στρατιωτικής και πολιτικής συνεργασίας ή στην στρατηγική παρουσίαση του ΝΑΤΟ θα είχε υποδέστερο λόγο, δηλαδή ότι το ΝΑΤΟ εστιάζεται στο στρατιωτικό σκέλος. Διάβασα όμως ε, σχόλια πρώην διοικητών του ΝΑΤΟ, ε, δεν θα σας πω τώρα πού ακριβώς τα διάβασα, όπου λέγεται ότι the comprehensive approach, δηλαδή ακριβώς αυτή η συνεργασία πολιτικού και στρατιωτικού σκέλους, είναι, ε, ε, είναι στο επίκεντρο της στρατηγικής του ΝΑΤΟ. Οπότε θα ήθελα να σχολιάσετε και να μου πείτε, ε, θεωρώ ότι αυτά ήταν αντιθετικά, αντιφατικά με αυτά που είπατε εσείς. Επίσης, εσείς τώρα αισθάνεστε ότι πρέπει στο το Βερολίνο ΣΥΝ να αξιολογηθεί περιοριστικά. Διότι εγώ νόμιζα ότι η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του ΝΑΤΟ στο Βερολίνο ΣΥΝ ε, είναι μια θετική παρουσίαση. Αυτό λοιπόν είναι επίσης ένα σχόλιο επί του οποίου θα ήθελα να έχω κάποια απάντηση ε, ε, όσον αφορά την ε, θεσμική γενική ανανέωση του ΝΑΤΟ μπορώ να σκεφτώ δύο τομείς αρχικός η αρχή της συνένεσης που ήταν μια πολύ βασική αρχή στο παρελθόν στο ΝΑΤΟ και σε σχέση με αυτό το γεγονός ότι αυτό που δεν, ε, ε, τα κράτη που δεν συμμετέχουν σε μία εμπλοκή του ΝΑΤΟ δεν έχουν δικαίωμα να, να ακούγεται η γνώμη τους. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι για μικρές χώρες του ΝΑΤΟ ότι δεν έχουν δικαίωμα ε, διαβούλευσης και δεύτερον ότι συγχρόνως όμως πρέπει να συμμετέχουν συμμετάσχουν στα έξοδα. Και σε αυτό το κοινοβούλιο με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ε, ε, ξέρω πώς αξιολογείται τη γνώμη των μικρών κρατών. Και ε, τέλος ε, στις ερωτήσεις μου θα, ή στο σχόλιο μου θα ήθελα να σας πω ότι θεώρησα ότι ήταν πολύ καλό ότι μας ενημερώσατε και εύχομαι στο μέλλον ε, η διαδικασία στρατηγικής προ, στρατηγικού προγραμματισμού του ΝΑΤΟ να είναι πιο δημοκρατικός και διαφανής και να συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυρία Λούνασεκ σας ευχαριστώ για αυτή την εκτενή παρουσίαση διότι για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρον να σας ακούσω για πρώτη φορά. Υπάρχουν δύο θέματα που θα ήθελα να σας ρωτήσω. Αφενός για το Αφγανιστάν. Είπατε ότι η διέξοδος από το Αφγανιστάν απαιτεί πολύ περισσότερους πόρους αν σας κατάλαβα καλά. Στις τελευταίες εβδομάδες και μήνες συζητήθηκε σε διάφορα μέσα ενημέρωσης και γύρω από τον Ομπάμα και στις νέες χώρες ακούσαμε ότι ίσως είναι αναγκαίο να αποσυρθούμε ε, το, διότι δεν θα κερδίσουμε. Μέσα στο ΝΑΤΟ λοιπόν γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Δηλαδή ότι ίσως το Αφγανιστάν ε, δεν μπορεί να επιτύχει ε, όπως στην αρχή υποθέταμε και ότι το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να αποσυρθεί ε, σύντομα ε, διότι υπάρχει και η ε, δημόσια γνώμη η οποία επηρεάζει την στήριξη στον Ομπάμα επ' αυτού. Πιστεύω ότι πρέπει να αποσυρθούμε αλλά πιστεύω θα πρέπει να συζητήσουμε τι στρατηγική θα ακολουθήσουμε και ότι ίσως δεν θα πρέπει πλέον να στηρίξουμε την ε, οικονομική και ε, στρατιωτική συμμετοχή. Εσείς είπατε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και περισσότερο από αυτές που περιγράψατε, αλλά εγώ προέρχομαι από μία ουδέτερη χώρα, έχουμε ουδέτερες ε, και όχι ε, ενάντια στο ΝΑΤΟ γιατί η Αυστρία συμμετέχει στην, ε, ε, στην σχέση για την ειρήνη αλλά ορισμένοι είπαν ότι το ΝΑΤΟ απλώς συνενώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ΗΠΑ ενώ εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε επίσης να πιεστεί για να συμβάλλει στην πρόληψη μέσω ίσως της συνθήκης της Λισαβόνας η οποία δίνει περισσότερες δικαιοδοσίες στην εξωτερική πολιτική. Αυτά ήθελα να πω εδώ ε, διότι βλέπω ότι είναι κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ και που πιστεύουν ότι μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη και αν αυτή τη στιγμή έχουμε καλή συνεργασία. Ο κύριος Γκαλτιέρη. Και εγώ ε, ευχαριστώ τον Διευθυντή για την εξαιρετική του εισαγωγή και για τα θέματα τα οποία παρουσίασε και τα οποία έχουμε περιγράψει και μας, μας ενδιαφέρουν διότι θα έπρεπε να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο. Ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στο σημαντικό ζήτημα που αναφέρατε για την inside castle, outside castle άμυνα. Ιδιαίτερα την πυραυλική άμυνα. Και ακόμα πιο ιδιαίτερα το νέο πρόγραμμα της Αμερικανικής κυβέρνησης στην συζήτηση, στην ομιλία του στη Μόσχα, ο κ. Ράσμουσεν μίλησε για το ενδεχόμενο ρόλου της Ρωσία στο ΝΑΤΟ στον τομέα αυτό. Το άρθρο του Gates του New York Times έδειχνε ένα αρκετά σαφώς οριοθετημένο σχέδιο αμερικανικής προέλευσης κατά βάση. Ήθελα να ξέρω κάτι περισσότερο για το ρόλο του ΝΑΤΟ και το μέλλον του νέου αυτού προγράμματος. Μια πιο γενική ερώτηση επίσης για το θέμα της πυρηνικής αποτροπής στα πλέ και της σχετικής στρατηγικής του ΝΑΤΟ εν ώψη του τέλους του κόσμου και για να συνδέσουμε την πρώτη με τη δεύτερη ερώτηση ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με την με μια παράλληλη στρατηγική σε σχέση με την στρατηγική την αντιπυραυλική στρατηγική, μια συμφωνία που, στην οποία θα μετέχουν και οι δύο βασικές δυνάμεις ε, ε, που έχουν πυράβλους μεσαίου βελνικούς. Ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση ή ε, έχω να κάνω μία παρατήρηση διότι μέχρι τώρα έχω δει τον κύριο Διευθυντή μόνο στην ε, ε, τηλεόραση και μάλιστα επανειλημμένος ε, σύντομα και χάρηκα πολύ που άκουσα τώρα μια εκτενή παρουσίαση που ήταν ε, ε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχω μια ερώτηση σχετικά με ένα θέμα που είπατε ότι το μπούμεραγκ επανέρχεται πάντοτε στις συζητήσεις, δηλαδή οι σχέσεις με τη Ρωσία. Οι σχέσεις με τη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σχέσεις με τη Ρωσία και το ΝΑΤΟ ε, εγώ εκπροσωπώ την, ε, το κόμμα του Πρωθυπουργού ΤΑΣΚ και έχουμε κάνει πολλά για την βελτίωση των σχέσεων και αυτό το διευκρινίζω για να μην με θεωρήσει κανείς ε, αντιρωσικό αντίθετο προς τη Ρωσία. Αλλά ε, σχετικά με αυτό που ελέγχθη ε, από το ΝΑΤΟ και από τον πρόεδρο Ομπάμα για συνεργασία με τη Ρωσία είναι θέματα τα οποία κατανοώ. Ε, το ερώτημά μου είναι απλούστατα στις αναλύσεις σας για το ΝΑΤΟ. Λαμβάνετε υπόψη ότι τα κράτη-μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ενότητας και του ΝΑΤΟ είναι πρόθυμα ε, για συνεργασία. Εσείς αναρωτιέστε αν θέλει και η Ρωσία να συνεργαστεί τίθεται αυτό το ερώτημα διότι ε, το, η Ρωσία έχει πυράβλους στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ε, χθες ε, έγινε πάλι μία άσκηση στη, σε ρωσικό έδαφος και ε, η Ρωσία ε, ήθελε να προσωμιάσει ε, μία πολωνική επίθεση στην Λευκορωσία και η Ρωσία θα έτρεχε να συνδράμει την χώρα στην οποία είχαμε επιτεθεί. Είναι δυνατόν λοιπόν να έχουμε συνεργασία στρατηγική με, μέσα στον Άτομο μια τέτοια χώρα αυτή η χώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. είναι ε, κατανοικό διότι εφόσον ε, είστε καλός προγραμματιστής είσαστε άλλωστε και το εκπρόσωπος ε, του ΝΑΤΟ, το φερέφωνο. Ήθελα λοιπόν να επανέλθω και εγώ στις σχέσεις με τη Ρωσία όπου αναφερθήκατε ή στα ενεργειακά ή την τρομοκρατία. Τι έχετε να πείτε για τον αφοπλισμό. Αυτό το θα ο πρόγραμμα που πρότεινε ο πρόεδρος Ομπάμα για έναν κόσμο χωρίς πυρηνική ενέργεια είναι κάτι ρεαλιστικό που είναι εφαρμόσιμο σύντομα ε, χωρίς πυρηνικά όπλα ε, ή, ή όχι. Επίσης ε, όσον αφορά τις σχέσεις του ΝΑΤΟ με τη Λευκορωσία. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζετε. Ευχαριστώ. Σας δίνω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω προφανώς να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές για τις ερωτήσεις τους και θα προσπαθήσω να απαντήσω χωρίς να ξεπεράσω το μήκος της προηγούμενης παρέμβασής μου, καταρχήν ε, ε, όσον αφορά την προσέγγιση Βερολίνο-Συν. Ίσως δεν υπήρξα όσο σαφής θα ήθελα και με συγχωρείτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία συνολική οργάνωση, το ίδιο συμβαίνει και με τον ΟΗΕ και λόγω της ποικιλομορφία τους έχουν στις ε, δομές τους στρατιωτικούς, δικαστές, αστυνομία, ε, ανθρωπιστική βοήθεια, διακυβέρνηση κτλ. Πράγμα το οποίο δεν σημαίνει ότι μπορούν να αναλάβουν όλες τις δουλειές μόνοι τους, αλλά θα πρέπει όλοι να συνεργαστούν. Παρ' όλα αυτά βέβαια μπορούν ε, να κάνουν ένα πακέτο μέσα στην οργάνωση και να έχουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση που δεν ισχύει στο ΝΑΤΟ διότι το ΝΑΤΟ δεν έχει πολιτικές ε, δυνατότητες παρόλο που για να απαντήσω σε μία ερώτηση εις, ε, την, ε, στο Αφγανιστάν το ΝΑΤΟ προσπαθεί να ανοικοδομήσει τις περιφέρειες αλλά προσωρινά μέχρι ότου μπορέσουν οι πολιτικές οργανώσεις να επέμβουν. Δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να παραμείνει επιμονή μου βάσεως και να αναλάβει πολιτικά καθήκοντα. Άρα προσπαθούμε απλώς να βοηθήσουμε τις άλλες οργανώσεις πολλές φορές και τις μη κυβερνητικέ ή τις επιχειρήσεις διότι αύριο θα μιλήσουμε ε, θα μιλήσω ο διευθυντή μου στο Λονδίνο με τι τις ασφάλειες για την αυτιλία, για την πειρατεία, για όλα αυτά. Δηλαδή η επιτυχία του ΝΑΤΟ δεν εξαρτάται μόνο από την στρατιωτική αποτελεσματικότητα διεξαγωγής των αποστολών, αλλά να μπορέσει να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΗΕ να αποδώσουν ίση σημασία μέσω του Αφγανιστάν και

και ε, να έχουν ε, τις ίδιες δυνατότητες διότι ε, διαφορετικά βλέπετε τι συμβαίνει δεν υπάρχει καμία ανοικοδόμηση ο πληθυσμός επιτόπου είναι όλο και πιο αποκαρδιωμένος και υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές. Το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει αποδεκτός σαν οργάνωση που συμμετέχει στο δίκτυο και να, μπορούμε να λογοθιόμαστε. Ε, επίσης, όσον αφορά το Βερολίνο ΣΥΝ, δεν έχω καμία αντίρρηση διότι δημιουργήθηκε στο Βερολίνο που είναι μια από τις αγαπημένες μου πόλεις. Ε, εάν όμως η Ευρώπη το χρησιμοποιήσει, αλλά στα 10 χρόνια της αμυντικής πολιτικής της η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οργανώσει 23 αποστολές εκ των οποίων μόνο δύο, μόνο δύο δηλαδή ένα πολύ μικρό ποσοστό ε, βασίστηκαν στο Βερολίνο ΣΥΝ. Ε, μία στο ΦΥΡΟΜ το 2001-2002 και στην Βοσνία που διατηρείται ακόμη. Η πραγματικότητα είναι ότι ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζονται είτε στη θάλασσα είτε στην Αφρικανική Ένωση ή στην Αντισαμπέμπα στο Κωσυφοπέδ με την αστυνομία Γιούλεξ ενώ δεν εφαρμόζεται το Βερολίνο ΣΥΝ. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την αστυνομία της ε, και τις δυνάμεις της Ιούλεξ. Ε, τι στρατηγική θα ακολουθήσουμε. Είναι χρήσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις που θέλει να το χρησιμοποιήσει σαν σύστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το Βερολίνο συν αποτελεί μάλλον εξαίρεση παρά κανόνα. Και έρχομαι τώρα στην ε, ερώτηση του Μάικελ, εάν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στρατιωτικές δυνατότητες. Ε, μας ε, έχει ζητηθεί να δανείσει το ΝΑΤΟ τις εγκαταστάσεις, το επιτελείο, τις δυνάμεις και εμείς προσφεθήκαμε διότι βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λέγεται ότι έχει αεροπλάνα, ναυτικές δυνάμεις, στρατιωτικές δυνάμεις, επιχειρησιακά ε, επιτελεία τα οποία δεν χρειάζεται ε, βάσει της ε, συμφωνίας Βερολίνο ΣΥΝ όπως χρειαζόταν ίσως στα μέσα της δεκαετίας του 90 όταν αναπτύχθηκε αυτή η ιδέα. Δεν, δεν λοιπόν η πραγματικότητα να προσαρμοστεί στην ιδέα αλλά μάλλον αντιστρόφων. Επίσης ένας ε, Γάλλος πρέσβης στο ΝΑΤΟ πριν μερικά χρόνια είχε πει ότι ε, ο στόχος Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν είναι να γίνει το πολιτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και είχε δίκιο. Δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να ε, διοικήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε να της δίνει εντολές. Τα δύο θεσμικά όργανα πρέπει να μείνουν τελείως ανεξάρτητα. Αυτό που θα θέλαμε όμως και ε, ε, θα ε, ψευδόμουν αν έλεγα κάτι διαφορετικό ήταν ότι θα χρειαζόταν μια στρατηγική αρμονία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τομείς που θεωρούμε ότι είναι ζωτικού ενδιαφέροντος και για τις δύο οργανώσεις. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν τα 22 κοινά μέλη και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο Αφγανιστάν παραδείγματο χάρη που είναι τόσο σημαντικά συμμαχία ώστε να αποτελεί μία περίπτωση ε, ιδιάζουσα ε, να μην έχουν τις ίδιες προτεραιότητες. Ε, όταν ήμουν με τον Γιάπτα Χιουσκέβα στο Λονδίνο ε, και συναντούσαμε τον Τόνι Μπλε πριν από μερικά χρόνια, δεν είναι πολύ πρόσφατο, ήταν πριν μερικά χρόνια που ήταν ακόμη Πρωθυπουργό ο Τόνι Μπλερ. Ο Γιάψη λοιπόν του είχε πει, κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε συζητήσει ποτέ το Αφγανιστάν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ο Μπλερ είχε πει όχι. Και το ΝΑΤΟ ήταν ήδη στο Αφγανιστάν επί σειρά ετών τότε. Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ ευγνώμονες στη Σουηδική Προεδρία για τις προσπάθειές της να καταρτήσει μία αυγανική στρατηγική και να αναθεωρήσει τις θέσεις της ε, δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να διατάξει και να προδιαγράψει τι θα κάνετε. Υπάρχουν ε, περιπτώσεις που το ΝΑΤΟ μπορεί να κινηθεί μόνο του. Πολλές ε, αποστολές Ευρωπαϊκής Ενώσεως όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κινηθεί μόνη της αλλά και πολλές στρατηγικές περιπτώσεις που προσφέρονται για συνεργασία όπως τα Βαλκάνια όπου έχουμε παράλληλες συμπληρωματικές διαδικασίες. Αν κοιτάξουμε όμως άλλους τομείς βασικούς για την ασφάλειά μας όπου απειλείται και η Ευρώπη και η Αμερική από μία αποτυχία χρειάζεται στρατηγική συνεργασία. Προφανώς όμως ε, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει το πολιτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Το νέο ΝΑΤΟ όμως δεν μπορεί να παρακολουθεί απλώς εκλογές ή να εκπαιδεύει η αστυνομία χωρίς να χρειάζεται κανείς να ντρέπεται που χρειάζεται να εμπλακεί σε μια τέτοια δραστηριότητα. Λοιπόν, όσον αφορά το εάν θα έπρεπε να συζητήσουμε με τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Βε, βεβαίως δεν κρύβουμε ότι καλό θα ήταν να υπάρξει διεύρυνση. Πρέπει να εξηγήσουμε στην Ρωσία γιατί θεωρούμε ότι οι χώρες αυτές έχουν τον όνειμο δικαίωμα να προσχωρήσουν στον ΝΑΤΟ εάν καλύψουν τα κριτήρια του ο ΑΣΕ και επίσης να αντιληφθούμε ε, γιατί η Ρωσία θεωρεί ότι θα απειληθεί από μια διεύρυνση του ΝΑΤΟ ή από τα πυρηνικά όπλα του ΝΑΤΟ σε ε, ε, ορισμένα κράτη-μέλη. Πρέπει όμως συγχρόνως να είμαστε διάφανοι για το τι κάνουμε στην Ουκρανία και στη Γεωργία για να μην δώνουμε τον εντύπωση ότι κινούμαστε πίσω από την πλάτη τους. Ε, θα πρέπει να είναι σαφές αυτό. Όσον αφορά ε, ε, τους οικονομικούς πόρους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενώσης το κάλυψα οι συμμαχίες. στο κολέγιο μου της Οξφόρδης υπάρχει ένα έμβλημα ad hoc is a mockery. Δηλαδή είναι αστείο να μιλάει κανείς για εστιασμένες δράσεις, Παραδείγματο χάρη οι περιοχές. Γιατί λοιπόν υπάρχουν χώρες σαν τη Νέα Ζηλανδία οι οποίες θέλουν να συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ, διότι γνωρίζουν ότι μπορούν να υποφεληθούν σε διάφορες περιπτώσεις από ιατρική βοήθεια, από δυνατότητα κενών Ω προσωπικού ότι υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες στο ΝΑΤΟ όπου διασφαλίζει στις διάφορες χώρες ότι μπορούν να βοηθηθούν από την συμμαχία είναι ε, ε, ε, πιο δύσκολο παραδείγματο χάρη να πει κανείς στο ΝΑΤΟ ότι αποχωρεί από ότι είναι από μια απλή συμμαχία. Ε, επιτυχία ή αποτυχία στο Αφγανιστάν. Δεν θα σας έλεγα ότι εάν αποτύχουμε στο Αφγανιστάν θα καταρρεύσει το ΝΑΤΟ, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Νέισβα ε, των θεσμών και ε, γι' αυτό χρειαζόμαστε το ΝΑΤΟ και για άλλα πράγματα, όχι μόνο για το Αφγανιστάν, για να ανταποκριθεί σε πολλές άλλες προκλήσεις και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η πρόκληση για το ΝΑΤΟ είναι ότι το Αφγανιστάν είναι μια πολύ απαιτητική αποστολή η οποία καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του χρόνου και των δυνάμεων και θα πρέπει να υπάρχει και πολιτική διαβούλευση για τα, τις άλλες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά τις μικρές χώρες. Στο ΝΑΤΟ έχουν μια φωνή την οποία δεν θα είχαν προς τις Ηνωμένε Πολιτείε ή τους μεγαλύτερους εταίρους. Νομίζω ότι ε, για τον ίδιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εφεκτική για τις μικρές χώρες ε, διότι οι μεγάλες χώρες συμβάλλουν στο να αυξηθεί το ανάστημα των μικρών και ε, ε, οι μεγάλες χώρες είτε συμμετέχουν σε οργανώσεις είτε όχι θα παραμείνουν μεγάλες, είναι νομιμοποιημένες ενώ οι μικρές νομιμοποιούνται μέσω αυτών και εάν υπάρχουν πολλές χώρες ε, που στηρίζουν μία πρόταση θεωρείται πιο βαρύνουσα. Το πιο βασικό όμω στοιχείο είναι να έχουμε αυτή την διάκριση μεταξύ της αποστολές σύμφωνα με το άρθρο 5 και τις οικειοθελείς αποστολές που δεν συγκαταλέγονται στο άρθρο 5. Ε, κανείς δεν θέλει να πάει στο Αφγανιστάν γιατί δεν είναι ε, αποστολή του άρθρου 5 η οποία όμως παραμένει σημαντική για το ΝΑΤΟ υπάρχουν ανθρωπιστικές αποστολές στενά συνδεδεμένες με την ασφάλεια όπου χρειαζόμαστε περισσότερη ε, ασφάλεια και όπως είπε ο Ρόμπερ Γκέις δεν μπορούμε να έχουμε ε, μία συμμαχία δύο επιπέδων. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς πολιτικά θα ε, διασφαλίσουμε την ίδια αλληλεγγύη στις επιχειρήσεις που δεν συγκαταλάγονται στο άνθρωπο 5 με αυτές που συγκαταλάγονται λέγονται στο άρθρο 5 διότι τα οικονομικά δεν μπορεί να αποτρέψουν από μία συμμετοχή διότι το 2006 έγινε ένα σεισμό στο Κασμίρ, θα το θυμάστε όλοι. Το ΝΑΤΟ αποφάσισε να στείλει μία αποστολή στο Κασμίρ, ουσιαστικά Ισπανούς μηχανικούς οι οποίοι πήγαν στο Κασμίρ, γύρισαν και ε, μετά είπε ο πρέσβης τους ευχαριστούμε ΝΑΤΟ αλλά αυτό μας κόστισε 25 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή εφόσον το ΝΑΤΟ αποφάσισε και διέταξε θα μας πληρώσει πληρώσετε και τότε είπε όχι, ε, η σειρά σας ήταν όταν ξεκίνησε η αποστολή και γι' αυτό την αναλάβατε εσείς. Ε, ε, έχουμε λοιπόν μία περίπτωση διεξαγωγής επιχειρήσεων με ρωσική ρουλέτα. Αν είστε εθελοντής θα τιμωρηθείτε, εάν δεν ε, προσφερθείτε δεν θα τιμωρηθείτε ή δεν θα φορολογηθείτε. Ε, βεβαίως κανείς δεν θα έκανε καμία προσπάθεια αν ε, ήξερε ότι κάποιος άλλος θα καλύψει τα έξοδα. Αλλά για τις κοινέ αποστολές που αφασίζονται από το ΝΑΤΟ όπου δεν μπορείτε να προβλέψετε κάτι όπως ένα ένας ή ε, ε, άλλη φυσική καταστροφή πρέπει να έχουμε δυνατότητα χρηματοδοτήσεως διότι διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ότι οι χώρες δεν θα καλύψουν τις μάχημες ε, αποστολές του ΝΑΤΟ. Ο, ο, ο πόλεμος στο Αφγανιστάν μπορεί να καταλήξει σε νίκη δεν έχουμε καμία ιστορική ιστορικό δίδαγμα το οποίο λέγει ότι δεν μπορεί να προχωρήσουμε έξι. στο Αφγανιστάν όλοι ήθελαν να, να προχωρήσουμε έτσι εκεί και κανείς δεν θέλει πίσω τους Ταλιμπάν. Το βλέπουμε αλλά οι Αφγανοί είναι ανυπόμονη ε, και η κοινή γνώμη θέλει να δει το φως στο, ε, στο βάθος του τούνελ. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να διατυπώσουμε ένα πρόγραμμα και ε, να οργανώσουμε την αποστολή. Uh, Πρέπει να δούμε πώς θα καλύψουμε τις ε, δυνατότητες να δούμε το φως στο βάθος του τούνελ διότι σε πολλές χώρες υπάρχουν ε, κυβερνήσεις ε, οι οποίες ενημερώνουν το λαό και υπάρχει πιο θετική αντιμετώπιση. Χώρες σαν την Αυστρία το το ΝΑΤΟ είναι μια μεγάλη ομπρέλα όπου έχουμε διάφορα ε, επιμόρφωση, ασφάλεια και μάχη με ομάδες ε, και σε διάφορες χώρες ε, υπάρχουν ειρηνευτικές δυνάμεις όπως στην Αυστρία, στην Ελβετία, στη Σουηδία. Η Ελβετία δεν είναι ούτε, στον, ούτε στα Ηνωμένα έθνη ούτε στο ΝΑΤΟ αλλά συμμετέχει εδώ και χρόνια με σεμινάρια νομικά για αφοπλισμό η Γενέβη χρησιμοποιείται σαν χώρο συνεδριάσεων παντού και ε, υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες να μπορέσει κανείς ε, να προχωρήσει. Τώρα, όσον αφορά τους πυράβλους και την άμυνα, αν επιτύχουμε και δεν είναι προφανές να λύσουμε το πρόβλημα του πυρηνικού αφοπλισμού για χώρες όπως το Ιράν και άλλες, όλο και περισσότερες χώρες ε, θα έχουν θα έχουν πυράβλους με ε, διάφορες κεφαλές ε, ε, βαλσικές, βιολογικού πολέμου κτλ. Και στην Ευρώπη υπάρχουν πύραυλοι δεύτερης και τρίτης γενιάς και η Αμερική και η Ρωσία μιλούν ε, για την αναθεώρηση της συμφωνίας των πυράβλων μέσου βεληνικούς αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε τι είναι οι δυνατότητες και η διοίκηση Ομπάμα έχει επικεντρωθεί προς το παρόν εις ε, το ε, χαμηλό βεληνικές αλλά μην πιστεύετε ότι η κυβέρνηση αυτή θα πάψει να ερευνεί, ίσως δεν εγκατηθιστά, αλλά δεν θα ερευνεί τα συστήματα μακριού βαλινεκούς. Επίσης η Ρωσία είναι ευπρόσδεκτη και η απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης να, να μην εγκαταστήσει στην Πολωνία και στην Τσεχία κεφαλές ε, δεν αποτελεί μέρος της ισορροπίας του ψυχρού πολέμου αλλά της συνολικής συνεργασίας και αντί για μία εξίσωση ε, σε ε, μια παλιά ισορροπία Ανατολής Δύσεως όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας στην ομιλία του μπορούμε να βοηθήσουμε να διατυπώσουμε με τη Ρωσία μια κοινή προσέγγιση διότι ο κίνδυνος δεν προέρχεται από τη Ρωσία αλλά από αλλού και προς τη Ρωσία και προς εμάς. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία να εστιαστούμε στους πραγματικούς κινδύνους και ξέρετε ότι μετά τη Νέα Υόρκη και τη συνάντηση του Μετβέντεφ ε, με τον Ομπάμα ε, μπορούμε να προσπαθήσουμε να πείσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να πείσει την, το Ιράν να είναι πιο διάφανο προς τις προθέσεις του. Τώρα, όσον αφορά το όραμα, ήδη έχει δοθεί κάποια ιδέα. Δεν μπορούμε συνεχώς να τονίζουμε ότι χρειάζονται πυρηνικά όπλα για να υπάρξει ευξημένη ασφάλεια. Όπως το είπε ο, ο κύριος Ελμπαραντέη της ατομικής του Γραφείου Ατομική Ενεργείας στη Βιέννη ε, πρέπει να μειώσουμε το πυρηνικό δυναμικό και όπως είπε και ο κύριος Ομπάμα ο ε, αφοπλισμός από πυρηνικά όπλα είναι μακρινή προοπτική θα πρέπει καταρχήν να υπάρξει συμφωνία συνεργασία μεταξύ Αμερικής και της Ρωσίας ε, προτού κάποια από αυτές τις δύο χώρες εγκαταλείψουν όλες τις πυρηνικές τους δυνατότητες. Θα πρέπει να υπάρχει το σωστό περιβάλλον, ασφαλεία, εμπιστοσύνης, όπου δεν θα χρειάζονται πλέον αυτά τα όπλα. Δεν μπορώ βέβαια να απαντήσω πλήρως. Δηλαδή τι ρόλο μπορεί να παίξει το ΝΑΤΟ σε αυτό το θέμα. Το αν η Ρωσία είναι έτοιμη ή πρόθυμη να συνεργαστεί με εμάς δεν το ξέρω. Εμείς πάντως είμαστε. Για την Πελαρούς έχουμε σχέσεις με την Πελαρούς η οποία μάλιστα πρόσφατα έδειξε μεγαλύτερη διάθεση να συνεργαστεί με το ΝΑΤΟ. Ιδιαίτερα για τη διαμετακόμιση προμηθειών προς το Αφγανιστάν. Μπορεί να ακούγεται περίεργος δρόμος για το Αφγανιστάν, αλλά υπάρχει. Βέβαια, αν η Μπελαρούς συμμερίζονταν τις αξίες μας θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι θέλει να πλησιάσει τον ΝΑΤΟ. Αν δείξει τέτοιο ενδιαφέρον θα ανταποκριθούμε. Δεν ξέρω αν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις, ελπίζω όμως. Ναι, νομίζω ήσασταν πληρέστατος. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας και για τις απαντήσεις σας. Ελπίζω να ξανασυναντηθούμε σύντομα όπως έχει κανονιστεί. Ευχαριστώ και εγώ για την υποδοχή σας. La réunion euh, terminée pour aujourd'hui. Η κανονική συνεδρίαση τελείωσε, αλλά έχουμε τους συντονιστάς, εάν θέλετε.